και ψηφίζουμε για το φάκελο, για το θέμα αυτό, στην Επιτροπή Ένβη στις 20 Μαρτίου. Οι συντονιστέ επίση αποφάσισαν να ξεκινήσει η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών για την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις κοινές, για τους κοινούς κανόνες εναρμόνισης δεν έχει ακόμα οριστεί συγκητή από την Επιτροπή μα. Θα ανοίξει η προθεσμία για τι τροπολογίε στην Επιτροπή μα και μετά θα ψηφιστεί στην ΕΛΒΗ η έκθεση. Η διαδικασία είναι ίδια με την προηγούμενη που σα περιέγραψα. Αυτή τη φορά η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή είναι η Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη Ρέτζι. Η προθεσμία λοιπόν για την υποβολή τροπολογιών είναι 6 Μαρτίου στι 11 το πρωί πάλι και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή ΕΝΒΗ στι 25 και 26 Απριλίου του 2018. Για τη σημερινή συνεδρίαση έχουμε 21 γλώσσες, ε, διερμηνία από δηλαδή και ως συνήθως τα έγγραφα διατίθενται ηλεκτρονικά από τη γνωστή εφαρμογή. Η συνεδρίαση μας θα μεταδοθεί στο διαδίκτυο. Περνάμε τώρα στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 105 του κανονισμού. Βασικά στοιχεία των συμβάσεων αποθήκευση δεδομένων που συνάπτονται στο πλαίσιο του συστήματος ίχνηλασιμότητας για τα προϊόντα καπνού. Ο κύριος Ομαρζέ είναι ο εισηγητής για το θέμα αυτό και θα εξετάσουμε το σχέδιο ψηφίσματος. Το λόγο θα λάβει πρώτος βεβαίω. ο εισηγητή, ο κύριος Ομαζέ. Έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Η συζήτηση αυτή είναι αναμενόμενη. Αφορά ένα σημαντικό ζήτημα της καταπολέμησης του καπνίσματος της αντιμετώπισης της παράνομου εμπορίου των προϊόντων καπνού και αφορά το σύστημα επαρκούς παρακολούθησης και ειχνηλασιμότητας για τα προϊόντα αυτά. Εννοείται ότι μπορεί να γίνει στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής μας επιτροπής η συζήτηση αυτή, παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα στο πλαίσιο της διαφάνειας, αλλά και με τρόπο αντιφατικό. Σε αυτή την Επιτροπή πρέπει να πραγματοποιηθεί η συζήτηση και όχι πίσω από κλειστές πόρτες, <clears throat> όπου ακούγονται καλά λόγια για να επηρεάσουν τις θέσεις που θα πρέπει να πάρουν αύριο οι βουλευτές. Όσοι ασχολούνται με την αντιμετώπιση του καπνίσματος και της βλάβες που προκαλεί στην υγεία, το θέμα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ιχνηλασιμότητα δεν είναι ε, στεγανό και δεν είναι ανεξάρτητο από τον κλάδο του καπνού. Οι καθηγητήριες γραμμές του 2008 που ενέκρινε η διάσκεψη των, των ε, ομάδων των ε, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κατά του καπνίσματος είναι ξεκάθαρες. Είναι απαραίτητο οι δημόσιες αρχές να προστατεύουν τη διαδικασία της σύλληψης και της υλοποίησης πολιτικών δημόσιας υγείας στην πολιτική κατά του καπνίσματος της καπνοβιομηχανίας όσο αυτό είναι δυνατόν. Η αδηγία που ονομάζεται του 2014 δεν έχει υλοποιηθεί ε, από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τήρηση αυτού του πλαισίου. Και ακριβώς σε αυτή την οδηγία υπάρχουν πολλές διατάξεις που αναθέτουν στην καπνοβιομηχανία διάφορες ευθύνες στο πλαίσιο του συστήματος παρακολούθησης και εχνηλασιμότητας προϊόντων καπνού που περιλαμβάνονται στην εκτελεστική πράξη που είναι υποσυζήτηση σήμερα. Επιπλέον, το άρθρο 8 του πρωτοκόλλου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προβλέπει ότι κάθε μέρος έχει την υποχρέωση να υλοποιήσει και παραθέτω πάλι ένα σύστημα παρακολούθησης και ειχνηλασιμότητας όλων των προϊόντων καπνού που ε, παρασκευάζονται ή εισάγονται στο εδαφός του και ότι κάθε μέρος δεσμεύεται να υλοποιήσει την παρακολούθηση και την ηχηλασιμότητα των προϊόντων καπνού, ώστε οι αρμόδιες αρχές του, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο καθεστώς παρακολούθησης και ηχνηλασιμότητας, να μην έχουν σχέση με την καπνοβιομηχανία και αυτούς που εκπροσωπούν τα συμφέροντά της, παρά μόνο στο βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητο. Η εκτελεστική πράξη που είναι υποσυζήτηση, όπως ή κατά πράξη, όπως και η συνδεδεμένη με αυτή η εκτελεστική πράξη, κατά τη γνώμη μου δεν τηρεί αυτές τις αρχές. Το σύστημα παρακολούθησης και εχνηλασιμότητας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, δεν ελέγχεται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Και οι σχέσεις που δημιουργούνται με την καπνοβιομηχανία ξεπερνούν αυτό που θα έπρεπε να είναι το απολύτως απαραίτητο. Στο, στην κατεξουσιοδότηση πλάξη ανατίθεται στην καπνοβιομηχανία να έρθει σε επαφή με αυτούς οι οποίοι έχουν συμβάσεις αποθήκευσης για να τους ε, προμηθεύσει τα ε, τα, δεδομένα για, τον, ε, για τα τσιγάρα. Είναι λοιπόν δεν είναι απίθανο ότι υπάρχουν υποψίες για, τις, για τους φορείς αυτούς. Και δεν το λέω εγώ. Υπάρχουν υποψίες ότι συμμετέχουν στην παράνομη διακίνηση τσιγάρων. Πρέπει να πω ότι τα μέλη της σύμβασης, τα μέλη της σύμβασης από καιρό έχουν αναγνωρίσει και παραθέτω και πάλι ότι η πολυμορφία των στρατηγικών και των τακτικών της καπνοβιομηχανίας που μπορεί, είναι πολλές γιατί προσπαθεί να παρέμβει στα μέτρα αντιμετώπισης του καπνίσματος. Και για μας αυτό συνεχίζεται μέσω αυτής της ε, κατεξουσιοδότηση πράξης και των, ε, εφαρμοστικών πράξεων, των εκτελεστικών πράξεων που είναι ε, συνδεδεμένες με αυτές, Είναι δυνατόν να προταθούν βελτιώσεις με το πώς έχουν τα, σε σχέση με το πώς έχουν τώρα τα πράγματα. Αλλά δεν μπορούμε και να πούμε ότι το σύνολο των σχέσεων μεταξύ των κρατικών αρχών και της καπνοβιομηχανίας θα διαραγούν από το σύστημα παρακολούθησης και εχνηλασιμότητας που προτείνεται σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και δεν είμαι σε θέση να καταλάβω πώς, όπως δεν θα καταλάβουν και οι Ευρωπαίοι πολίτες, ότι για να λειτουργήσει μία επιλογή μεταξύ πολλών συστημάτων, από το πλέον ανεξάρτητο από την καπνοβιομηχανία μέχρι το λιγότερο ανεξάρτητο, το βασικό κριτήριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να είναι η αποτελεσματικότητα όσον αφορά το κόστος για την καπνοβιομηχανία. Προσωπικά θεωρώ ότι όσον αφορά τη δημόσια υγεία και κυρίως όταν πρόκειται για αντιμετώπιση του καπνίσματος πιο σημαντικό είναι για την Επιτροπή να σκέφτεται υπό την έννοια του ωφέλους για την ανθρώπινη υγεία και όχι στο όνομα κάποιες αποδοτικότητας κάποιου κόστους της καπνοβιομηχανίας. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν καταθέτω την ε, αντίρρηση αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι δεν υπάρχει πλέον κανένα περιθώριο ελιγμών και ότι πρέπει να δεχτούμε το κείμενο ως έχει. Πολύ καλά. Τι σημαίνει όμως αυτό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι σημαίνει η κοινοβουλευτική δημοκρατία για την Κομισιόν και θέτω το ερώτημα. Δεν έχουμε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή άλλη επιλογή παρά μόνο να αποδεχτούμε και δεν έχουμε λόγο παρά μόνο το μόνο που μπορούμε να κάνουμε να πούμε ότι όλα είναι εντάξει τότε δεν έχουμε καμία χρησιμότητα. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωση του Κοινοβουλίου, είναι καθήκον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής μας του περιβάλλοντος να μην κάνει δίκες προθέσεων, αλλά να ζητά από την Κομισιόν να εργάζεται και να κάνει βελτιώσεις όταν θεωρούμε ότι η πράξη που μας προτείνει είναι προβληματική είναι, θα ήταν είναι ανεύθυνο από πλευρά της Κομισιόν να μας απαντά ότι τελικά αυτή η πράξη είναι, σε αυτή την πράξη μπορούμε να πούμε είναι ή όχι. Αυτά είναι περίπου τα ίδια, παραδείγμα, τα ίδια ε, επιχειρήματα με το γλυφοσάτ, με τους ε, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και μια σειρά από άλλα θέματα. Όλοι ξέρουν, Όλοι λένε οι ε, πολίτες κάνουν λάθος, λάθος η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας κάνει λάθος, οι επιστήμονες κάνουν λάθος, οι πάντες κάνουν λάθος εκτός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καλό τους συναδέλφους να έχουν αύριο το θάρρος και την δύναμη που έχει ανατεθεί στο κοινοβούλιο μας να υπερψηφίσουν την αντίρρηση που έχω καταθέσει μόνο έχοντας κατά νου την ανθρώπινη υγεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μαζιζέ. Και τώρα ο λόγος στους και εισηγητές. Ο κύριος Φλόρενς πρώτος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, σας συμπαθώ πάρα πολύ. Είσαστε πολύ ταλαντούχος. Και δεν το λέω ε, τυχαία. Ο... Η κυρία Μακάβαν και άλλοι Γάλλοι συνάδελφοι ε, πολέμησαν πολύ σκληρά για τα προϊόντα καπνού για να περιοριστούν ε, και αυτό που πετύχαμε δεν είναι ε, λίγο. Δεν θέλω βεβαίως να εγκομιάσω τα όσα έγιναν ως τώρα απλώς, αλλά πραγματικά και οι σοσιαλιστές με όσα έκανε η Λίντα Μακάβαν ήταν αρκετά ικανοποιημένοι. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι έχετε κάποια καθυστέρηση. Αυτή η χνασιμότητα που προβλέπετε δεν σας αρέσει τώρα, όμως έπρεπε η πολιτική σας οικογένεια να έχει πάρει μέρος στους τρισμερείς διαλόγους πολύ εγκαιρότερα και να έχει λάβει μια πιο ε, αποφασιστική θέση στα πράγματα. Έρχεστε λιγάκι εδώ σαν τους χωροφύλακες της Όφενμπαχ. Και με αυτό το έγγραφο πραγματικά δεν θα καταφέρουμε ούτε ε, κατά ένα βήμα να μετακινήσουμε τα πράγματα. Πρέπει να γίνει κάτι πιο δραστικό. Συζητούμε πολύ την ανεξαρτησία. Ποιος είναι ανεξάρτητος ε, Είμαι σε θέση σε κάποια ερωτήματα να απαντήσω ως ανεξάρτητος και σε κάποια άλλα όχι. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να ληφθούν οριστικές αποφάσεις εδώ. Η Επιτροπή μας ε, για την λήψη αυτών των μέτρων εργάστηκε πάρα πολύ καλά και θέλω να το υπογραμμίσω. Και με όλα τα κοινοβουλευτικά μέσα που έχω στη διάθεσή μου θα ε, φροντίσω αυτή η αντίρρηση, η ένσταση να μην τύχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αυτό ήθελα να πω. Ε, δεν έχω τίποτα εναντίον σα, αλλά θα σα έλεγα να βρείτε κάποιο άλλο θέμα για να προβάλλετε αντίρρηση όπου να έχετε μεγαλύτερη επιτυχία. Πρόεδρο. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριο Πανιού. Πρόεδρε, συνάδελφοι, να πω ότι πρόκειται για ένα θέμα που το γνωρίζουμε καλά εδώ στην Επιτροπή ΕΝΔΙ. Το είπε τώρα και ο κύριος Φλόρενς. Η δουλειά που κάναμε υπό την αιγίδα της Λίντα Μακάβαν για να εγκριθεί επιτέλους μια οδηγία ε, καταπολεμώντας από πολιτικής άποψης αυτά που θέλαμε ε, ήταν σημαντικό και εγώ το 2014 προείδρευα ε, και κινητοποιούσα ε, μια ομάδα εργασίας κατά της, ε, του παρεμβατισμού της καπνοβιομηχανίας σε ό,τι έχει να κάνει με προϊόντα καπνού. Η αγωνιστικότητα που δείξαμε λοιπόν σε αυτή την ομάδα εργασία αντικατοπτρίζεται με όσα εγκρίθηκαν και έγινε και ένα άλλο αγώνα τον οποίο κερδίσαμε. κερδίσαμε λόγω χάρη με την χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη χρηματοδότηση που διεκόπη τη χρηματοδότηση προς τους καπνοβιομηχάνους λοιπόν. Ε, διεκόπη μια σύμβαση τον Ιούλιο που ήταν ε, πολύ παλιά ε, στην ηλικία. Είδαμε λοιπόν φέτος τον παρεμβατισμό της καπνοβιομηχανίας σε πολιτική, στις πολιτικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και αυτό το περιορίσαμε αρκετά στριμώχνοντας κάπω την καπνοβιομηχανία. Ο αγώνα όμω συνεχίζεται. Ο αγώνα συνεχίζεται και με την εχνηλασιμότητα. Και πρέπει να πω ότι αυτά που αποφασίσαμε στο πλαίσιο της οδηγίας του 2014 είναι ανεξάρτητη η χνηλασιμότητα. Η χνηλασιμότητα σε επίπεδο κρατών μελών που αυτά την διοργανώνουν, αυτά την διευθύνουν και να μην ε, αυταπατώμεθα τον πολιτικό αγώνα τον κερδίσαμε. Από το 2019 η χνηλασιμότητα θα είναι βεβλημένη. Δεν θα μπορεί να γλιτώσει κάποια μηχανία μέσα από τις κωδικοποίησεις. Δεν θα μπορεί να έχει πια το μονοπόλιο που θέλει. Τη χνηλασιμότητας δηλαδή. Όμως ταυτόχρονα άλλος αγώνας πρέπει να δώσουμε είναι το μονοπόλιο αυτό να μην αντικατασταθεί από ένα άλλο μονοπόλιο. Υπάρχουν επιχειρήσεις στην Ευρώπη που θέλουν να αντικαταστήσουν το κώδικα αυτό με άλλο σύστημα που να μην είναι ούτε διαφανές ούτε ανεξάρτητο. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε η κατεξισοδότηση πράξη να ε, σχεδιαστεί έτσι, ώστε να επιτρέψει όντως να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια. Διότι το γνωρίζουμε. Εάν αυτή η κατεξοσοδότηση πράξη και βάσει τον πολιτικό αγώνα του 2014 και των ε, περαιτέρω εξελίξεων, εκεί θα ε, έχουμε την ανεξαρτησία που θελήσαμε και όσα ε, ζητάει το άρθρο 105. Ε, συγγνώμη, όσα ζητάει ο κώδικας που έχει προβλεφθεί. Εδώ λοιπόν 2017 ε, ήταν η έγκριση του συστήματος και όχι 2016 και το 2022 θα φτάσουμε τις 40 μονάδες που θέλουμε σε σχέση με τις 35 που ισχύουν σήμερα. Βάσει της μελέτης λοιπόν του ΠΟΗ θα υπάρξει ε, ευνοϊκότερη μεταχείριση των εταιριών που έχουν ακολουθήσει τις ε, προδιαγραφές του από, το, από δεκαετία τώρα έχουν λάβει τα τεχνικά μέτρα που απαιτούνται για να σεβαστούν τι προδιαγραφέ του ΠΟΗ. αυτό τον αγώνα τον δώσαμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και τον κερδίσαμε. Ε, εν τέλει, και θα ολοκληρώσω, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να υπάρχει απαραίτητη επαγρύπνηση και η ανεξαρτησία καθώς και η ψηφοπιστία του συστήματος ίχνη να εξελιχθεί όπως θέλουμε. Οπότε ο εισηγητής μας ο κύριος Γιουνούς ο τον οποίο εκτιμώ καθόλου ως ε, βουλευτή στο έργο του, τώρα ανακαλύπτει το πρόβλημα ε, σε όλες του τη διαστάσεις, στο εύρος του πολιτικού αγώνα. Ε, αν είχατε έρθει στην ομάδα εργασία μα, θα είχαμε έναν παραπάνω στρατευμένο για να μα επιτρέψει να κερδίσουμε και άλλου αγώνε όπω αυτού που κερδίσαμε τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η, ο επόμενος ομιλητή η κυρία Γιατενμάκη. Αγαπητή Πρόεδρε, η κυρία είναι η Σκιώδης, αλλά μου ζήτησε να πάρω το λόγο εκ μέρους της, γιατί δεν κατάφερε να έρθει σήμερα το απόγευμα στη συνεδρίαση. Θέλει να υπογραμμίσει τα εξή σημεία. Το επιχείρημα που προβάλλει ο κύριος μαρζέ είναι αυτό που ακούσαμε από τα μέλη της ομάδας EFT πέρυσι τον τέλος Σεπτεμβρίου και η Επιτροπή τα, τα ε, απέρριψε με μεγάλη πλειοψηφία συμπεριλαμβανομένων και των μελών της ε, Άλντε. Η κυρία Βρύς θέλει να μας υπενθυμίσει ότι το προτινόμενο σύστημα παρακολούθησης και χνηλασιμότητας ε, αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο παράγονται τα τσιγάρα και καπνό για ε, τύλιγμα τσιγάρων θα υπάρχει θα υπό έλεγχο. Στην ουσία είναι εντελώς νέο το σύστημα. Οι μοναδικοί κωδικοί θα προκύπτουν από ένα, μια, έναν ανεξάρτητο τρίτο που όπου δεν θα έχει καθόλου η καπνοβιομηχανία εμπλοκή στο σχεδιασμό του συστήματος. Κυρία Βρύση επίσης αναφέρει ότι, ότι το νέο σύστημα εχνηλαστιμότητας δεν είναι τέλειο. Σαφώς υπάρχει περιθώριο περαιτέρω βελτίωσης δεδομένου ότι θα εξακολουθούν να έχουν ρόλο οι καπνοβιομηχανίες για τις, ε, στις εταιρείες συγκέντρωσης δεδομένων για την αποθήκευση. Όμως, αν και χρειάζονται πιο αυστηρά κριτήρια, πιστεύει ότι δεν υπάρχει εγγύηση ότι το σύστημα θα είναι εντελώς ανεξάρτητο από τις μεγάλες καπνοβιομηχανίες. Τέλος δε, η κυρία Βρύς θέλει να υπογραμμίσει ότι αν η αντίρρηση αυτή πραγματικά περάσει, δεν θα εφαρμοστεί ολόκληρο το σύστημα ε, παρακολούθησης και ειχνηλασιμότητας όπως έχει προγραμματιστεί το Μάιο του 19 και αυτό θα θεωρηθεί μεγάλη νίκη των καπνοβιομηχανιών. Και αυτό δεν νομίζω ότι είναι μήνυμα που θέλει να στείλει η Επιτροπή μας. Γι' αυτό συ, συστήνει η ομάδα Άλτε να καταψηφίσει την αντίρρηση αύριο το πρωί και να συνεχίσουμε να δίνουν εμπιστοσύνη στη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ στην ε, μάχη κατά των προϊόντων καπνού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα η κυρία Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, θα είμαι σύντομη. Από άποψη τώρα του ECR θεωρούμε ότι πρόκειται ακόμα για ένα θέμα όπου οι αντιρρήσεις ε, ε, θα βλάψουν περισσότερο από ό,τι θα ωφελήσουν παρά τις καλές προθέσεις. Μερικές φορές, κατά εξαίρεση, υπάρχουν περιπτώσεις που η νομοθεσία που έχει συμφωνηθεί με συναπόφαση πρέπει να εξεταστεί πριν τεθεί ισχύ, αλλά πραγματικά πρέπει να είναι εξαιρέσεις και στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι τέτοια περίπτωση. Συμφωνώ με την κυρία Βρύς ότι αν αυτό δεν το αφήσουμε να υλοποιηθεί, θα αφήσουμε όλο τον τομέα ανοιχτό προς εκμετάλλευση. Το σύστημα δεν θα μπορέσει να υλοποιηθεί πριν από το 2022, γιατί δεν θέλουμε να προκαλέσουμε καθυστέρηση. Ακόμα και αν το σύστημά μας δεν είναι τέλειο, υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπιστεί αυτό από την ώρα που θα δημιουργηθεί το σύστημα. Δεν ε, συμφωνώ ότι ακούσαμε κάποιο λόγο για να αλλάξουν αυτά ε, τώρα, εδώ και τώρα, και γι' αυτό ζητώ να καταψηφιστεί. Ευχαριστώ. Άλλο μέλος που θα ήθελα να πάρει το λόγο. Αν όχι, στρέφομαι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η... από τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ ο αντιπρόεδρος, Σα ε, ο ε, υποδιευθυντής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ που καλέσατε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, τοποθετηθεί για τα βασικά στοιχεία των συμβάσεων αποθήκευση δεδομένων που συνάπτονται στο πλαίσιο του συστήματο συνεκλασιμότητα για τα προϊόντα καπνού και τη σχετική κατεξουσιοδότηση πράξη, τον κανονισμό, η οποία εγκρίθη στι 15 Σεπτεμβρίου 2017 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ίδια μέρα και ο εκτελεστικό κανονισμό για το σύστημα εχνηλασιμότητα που θα ιδρυθεί και για τη σχετική εφαρμοστική απόφαση για τα στοιχεία ασφάλεια των προϊόντων καπνού. Από κοινού όλα αυτά τα μέτρα καθορίζουν τι βασικέ προποθέσει για τη δημιουργία και τη διαχείριση ενό ευρωπαϊκού συστήματο εχνηλασιμότητα και στοιχεία ασφάλεια για τα προϊόντα καπνού, Όπω προβλέπουν τα άρθρα 15 και 16 τη οδηγία για τα προϊόντα καπνού. Να ξεκινήσω επιβεβαιώνοντα ότι έχουμε σημειώσει με προσοχή τα στοιχεία του σχεδίου ψηφίσματο που σήμερα συζητάτε και θα ήθελα να πω γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι δεν είναι βάσιμες οι αμφιβολίες που εκφράζει το σχέδιο ψηφίσματος. Το θέμα διαδικασίας είναι σημαντικό, το διαδικαστικό δηλαδή. Ξέρουμε ότι οι περισσότερες αμφιβολίες που εκφράζει το κείμενο έχουν να κάνουν με πτυχές του συστήματος εχνηλασιμότητας που ε, τις ε, διευκρινίζει ο κανονισμός ε, και όχι ο κατεξουσιοδότης κανονισμός που τώρα ε, εξετάζεται. Θα πρέπει να θυμίσω ότι από τις 29 Σεπτεμβρίου 2017 η Επιτροπή ΕΝΒΗ ε, απέρριψε άλλη ένσταση κατά του κανονισμού αυτού και η σχετική συζήτηση έγινε στην Επιτροπή ΕΝΒΗ όπου είχε εκφραστεί η άποψη ότι δεν θα πρέπει να ε, εμποδιστεί από το να τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός. Ε, είναι σημαντικό ότι πολλά από τα, από τα θέματα που γύρονται στο κείμενο του ψηφίσματος πρέπει να τύχουν κάποιες απάντησεις το βασικότερο θέμα της ανεξαρτησίας του συστήματος εχνηλασιμότητας, ανεξαρτησίας από την καπνοβιομηχανία. Να βεβαιώσω τους ευρωβουλευτές ότι υπάρχουν πολλές ε, δικλείδες ασφαλείας που έχουν συμπεριληφθεί στον κανονισμό, ώστε το σύστημα να παραμείνει πλήρως υπό τον έλεγχο των Εθνικών Αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι λεπτομέρειες των ε, ε, δικλειδών αυτών ασφαλείας έχουν περιληφθεί στα δελτία ασφαλείας που ετοίμασαν οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή ΕΝΒΗ. Δύο όμως είναι μεγαλύτερε σημασία. Πρώτον, η συμπερίληψη ενό συνόλου αυστηρών και λεπτομερών στοιχείων ε, αποτίμηση για να είμαστε βέβαιοι ότι όλα τα τρίτα μέρη που εμπλέκονται σε αυτό το σύστημα, όπω και οι υπεργολάβοι, ε, είναι ανεξάρτητοι από την καπνοβιομηχανία. Ταυτόχρονα, αυτά τα λεπτομερή κριτήρια έχουν να κάνουν με την νομική ανεξαρτησία του, την οικονομική του και την απουσία συγκρούσεων συμφερόντων. Δεύτερον, να επισημάνω ότι ο συνολικός σχεδιασμός του συστήματος επιτρέπει στις αρχές να ελέγχουν το σύστημα αυτό. Ε, και ως προς το συγκεκριμένο σημείο ε, μιλάω για τον διορισμό της βασικής απόδοσης του καθήκοντος των βασικών επιθεωρητών στα κράτη-μέλη. Εκείνοι ορίζουν τρίτα μέρη, ε, πλήρως συμμορφούμενοι με τα κριτήρια ανεξαρτησίας, ώστε να αναλάβουν αυτό το ρόλο ή τέλος πάντων μπορούν να τον αναλάβουν και μόνοι τους να επιβεβαιώσω ότι αυτή η αρμοδιότητα προέκυψε ως η βασικότερη αρμοδιότητα στο σύστημα ελέγχου μετά από λεπτομερέστατη αποτίμηση που έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οδήγησε στην ε, ε, σύνταξη της πράξης αυτές, ε, αυτή η προετοιμασία έχει να κάνει με τεχνικές ε, συζητήσεις με ειδικούς και εμπειρογνώμονες, με εκπροσώπους των κρατών μελών και με εκπροσώπους των εταιριών. Ε, θεωρήσαμε ότι ο δερισμός σε άλλους φορείς ενός περιορισμένου συνόλου υποτεχνικών αρμοδιοτήτων, ώστε στα πακέτα λόγω χάρη να ανοιχνεύουν τα ειδικά στοιχεία ασφαλείας, αυτό δεν θα θέσει αμφιβόλο το όλο σύστημα ηχνηλασιμότητας, εφόσον υπάρχουν και άλλοι παράγοντες ελέγχου της ασφάλειας, όπως αυστηρότητα το σύνολο δεδομένων, στο οποίο τώρα θα έχουν πρόσβαση εγκαίρως οι κεντρικές αρχές. Γι' αυτό έχω την πεποίθηση ότι το σύστημα ασφαλεία και συνεργασιμότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πλήρω ανεξάρτητο από την καπνοβιομηχανία και υπό τον έλεγχο των εθνικών αρχών. Άρα θα είναι σε θέση να συμμορφωθεί πλήρω με τι απαιτήσει ε, του άρθρου 8 του πρωτοκόλλου FCTC. Ε, μερικά βασικά στοιχεία ε, των ε, του κανονισμού που συζητιούνται τώρα έχουν να κάνουν με τις προϋποθέσεις για τους καπνοβιομηχάνους και ε, τις συμβάσεις που συνάπτουν με ανεξάρτητα τρίτα μέρη καθώς και το πού θα γίνεται η αποθήκευση των δεδομένων. Όλες αυτές οι προποθέσει ορίζονται από την ίδια την οδηγία για τα προϊόντα καπνού, το άρθρο 15.8. Ε, ο κατεξουσιώδης κανονισμός απλώς αντικατοπτρίζει αυτές τις προποθέσει και διευκρινίζει ποιε είναι οι βασικές συμβασιακέ προποθέσει που πρέπει να γίνονται σεβαστέ. Να έχουμε κατά νου ότι αυτή η συμβασιακή σχέση θα έχει να κάνει με το κόστο τη αποθήκευση δεδομένων, το οποίο αναλαμβάνει η καπνοβιομηχανία. Κάτι το οποίο προβλέπεται σαφώ από, από το άρθρο 8 του πρωτοκόλλου FCTC. Για να ολοκληρώσω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τη άποψη ότι ο τη κανονισμό που τώρα συζητάτε και συνάδει με τι αρμοδότητε που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη βασική πράξη τη σχετική οδηγία δηλαδή και συμμορφώνεται πλήρω με την νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνή νομοθεσία, δηλαδή την ε, νομοθεσία για τα προϊόντα καπνού και την πρωτοκόλλο FCTC. Το να τροποποιηθεί ο κανονισμό αυτό βάσει των όσων ζητά τώρα το σχέδιο ψηφίσματο δεν θα πετούσε απλώ τροποποίηση των ήδη εγκεκριμένων εφαρμοστικών κανονισμών, αλλά θα ξανάνοιγε την όλη οδηγία για τα προϊόντα καπνού. Και αυτό θα είχε την αναπόφευκτη συνέπεια να καθυστερήσουμε σοβαρώ στην όλη όλη η ίδρυση του συστήματο και τη λειτουργία του. Άρα θα μπορούσε κάποια μηχανία να λειτουργεί ανεξέλεγκτα από την άποψη τη εγκλασιμότητας για το άμεσα προσεχές μέλλον. Αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να το αποφύγει με κάθε κόστο. Ευχαριστώ πολύ. πρόεδρο, σα ευχαριστώ. Έχετε να πείτε κάτι για ένα λεπτό, νομίζω, έτσι είναι. Α, κύριο Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Σε ένα λεπτό. Ένα λεπτό χρόνο αγορεύσεως. Να σας πω ότι εξής, είμαστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Και δίκαιο είναι των βουλευτών να προβάλλουν ενστάσεις και όταν το πράττουμε αυτό δίνουμε ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα στον ελεγκτικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το δικαίωμα λοιπόν αυτό το ασκούμε και είναι φυσιολογικό και δεν υπάρχει κανένας λόγος να ε, διεγείρεται κανείς. Βρίσκομαι σε μια κατάσταση κάπως ασυνήθη, μόνος έναντι όλων. Η ιστορία θα δείξει ποιος από εσά ή από εμά έχει τελικώς δίκιο. Και νομίζω ότι πολλοί από εσά λησμονείτε το σκάνδαλο τα σκάνδαλα της ε, καπνοβιομηχανίας και πολλοί ξεχνούν τις πιέσεις που ασκούνται. Θα πρέπει λοιπόν να εμπιστευτώ τον λόγο σας. Να θεωρήσω ότι δεν έχει ασκηθεί καμιά πίεση. Να θεωρήσω ότι δεν έχει χειραγωγήσει τις διάφορες ενώσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να θεωρήσω ότι δεν έχουν ασκηθεί πιέσεις επί των Ευρωβουλευτών. Καλώ, σα πιστεύω, πιστεύω τον λόγο σας, αλλά διαπιστώνω ότι κανείς δεν κατέθεσε αντίθετα επιχειρήματα και ότι οι βελτιώσεις πρέπει να επέλθουν. Και εγώ βασίστηκα και πιστέψτε με ότι έχω διαρκείς επαφές με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Και όλοι μου λένε ότι το άρθρο 8 δεν τηρείται και ότι οφείλουν να επέλθουν βελτιώσει. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Όλοι μπόρεσαν λοιπόν να τοποθετηθούν. Θα ψηφίσουμε αύριο. Θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα ψηφοφορία στην Επιτροπή μας και τον Μάρτιο στην Ολομέλεια θα είναι το η ψηφοφορία ε, επί του ψηφίσματος. Τώρα, ακολουθεί η γνωμοδότηση πρωτοβουλίας για τις σχέσεις με την Κίνα του εισηγητού κυρίου Στέφαν Εκ, στον οποίο παραδίδω τον λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα πρώτα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι η παρούσα Επιτροπή συζητεί την γνωμοδότηση για λογαριασμό της Επιτροπής Εξωτερικών για τις σχέσεις με την Κίνα. Θεωρώ ότι παρόλη την δικαιολογημένη κριτική και από πολίτες και από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων απέναντι στην Κίνα, η Ευρώπη έχει συμφέρον να συνεργαστεί για να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό της Κίνας, αλλά και να συνεργαστεί με τη μεγάλη αυτή χώρα για να δράσει σε τομείς όπως το περιβάλλον η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ζωτικό συμφέρον για την διατήρηση καθαρού του περιβάλλοντος και για την αφαίρεση του διοξιδίου του άνθρακος. Η Κίνα που είναι και ο μεγαλύτερος παραγωγός τροφίμων στον κόσμο έχει και την μεγάλη ευθύνη να προωθήσει τον αγώνα κατά της ε, ανθεκτικότητας στα αντιβιωτικά, γιατί είναι και ο μεγαλύτερος καταναλωτής τους. Τώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να βασιστεί σε άλλους για να ακολουθήσει μια αποτελεσματική περιβαλλοντική πολιτική, τώρα δεν ξέρω και αν ποτέ θελήσαμε να το κάνουμε αυτό, μας φαίνεται η Κίνα ως κατάλληλος εταίρος με τον οποίο σε συνεργασία η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αναλάβει ένα πρωτοποριακό ρόλο. Χωρίς την υποστήριξη των δύο μεγαλύτερων αυτών οικονομικών δυνάμεων του κόσμου, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί από μόνη της να κάνει πολλά πράγματα για την μετρίαση των ε, βαριών συνεπειών της αλλαγής του κλίματος, αύξηση του επίπεδου των θάλασσών, βαριές θεομηνίες και ούτω καθεξής. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να συνεργαστούμε πολύ στενά με την Κίνα για να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά τα προβλήματα που μόλις σας ανέφερα. Κίνα και Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται ήδη σε καλό δρόμο. Αν εξετάσουμε τις μεγάλες επενδύσεις που κάνει η Κίνα σε θέματα ηλεκτροκίνησης, καθώς επίσης και για την ηλιακή και ολική ενέργεια. Το 2016 οι κινέζικες επιχειρήσεις επένδυσαν 35 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη γνώμη μου, η περαιτέρω συνεργασία θα πρέπει να επεκταθεί στην έρευνα και στην επιστήμη και θα αποτελέσει έτσι μια καλή βάση για μια συνεργασία τεχνική, στη τεχνολογία, πρέπει να βρούμε τους καλύτερους τρόπους για να μειώσουμε στο ελάχιστο ή δυνατόν την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, του κλίματος και του ατμοσφαιρικού αέρα. Χρειάζεται ποιοτική ανάπτυξη και στην Κίνα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δοθούν περισσότερα κίνητρα για να δημιουργηθούν έτσι και εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης. Είμαι βέβαιος ότι θα βρει θετική απήχηση η γνωμοδότησή μου και με τον τρόπο αυτό θα δώσουμε και ένα πραγματικά θετικό και πολύ σημαντικό μήνυμα στις χώρες μας. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα, συνάδελφοι. Θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο κύριο Εκ για την έκθεση αυτή, για την κατάσταση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας, ιδίως ως προς τα περιβαλλοντικά θέματα. Θέλω να πω το εξή, κύριε Εκ. Πήγα στο βορρά της Νορβηγίας την περασμένη εβδομάδα. Στα σύνορα με τη Ρωσία, κοντά. Οι εκπρόσωποι των νορβηγικών αρχών μιλούσαν για επενδύσεις, για τις ανοιχτές πόρτες προς τη Ρωσία και λέγαν ε, έχουμε για κάτι προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ είναι να συνεχίσουμε τη συνεργασία, τους χρειαζόμαστε και ούτω καθεξής. Εγώ τους είπα δεν γίνεται αυτό, οι αξίες μας δεν μας το επιτρέπουν. Δεν μπορούμε να παραγωνίσουμε τις λεγόμενες core values, τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι και τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ξεχνάμε τους αγώνες ε, και τις προσπάθειες που έχουν γίνει. Είναι λοιπόν σημαντικό όντως στη σχέση μας με την Κίνα να θυμόμαστε και αυτή τη διάσταση ένα μέρο του είναι τα περιβαλλοντικά ζητήματα, αλλά υπάρχουν και τα ανθρώπινα δικαιώματα που είναι αλληλένδετα με τα περιβαλλοντικά, είτε αμέσω είτε εμέσω. Ξέρουμε τι γίνεται με το θέμα της περιβαλλοντικής μετανάστευση, Ένα ζήτημα που ε, στην Κίνα έχει σαφώς ε, μια ιδιαίτερη διάσταση, αλλά και το θέμα των πολιτικών ελευθεριών στην ε, Κίνα. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Πάντω να πω ότι σε σχέση με το κείμενό σας, Ευτυχώ καλύπτεται ένα πολύ μεγάλο μέρο των ζητημάτων που είναι σοβαρά, που ε, άπτονται των περιβαλλοντικών ε, μεριμνών μα. Πιστεύω ότι το κείμενο μπορεί να βελτιωθεί και για να βελτιωθεί καλό θα ήταν να λάβει υπόψη και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτό λοιπόν θα υποβάλω κάποιε τροπολογίε στο αρχικό κείμενο, διότι δεν μπορούμε να παραβλέπουμε τις διαρκείς παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα. Είτε με, αμέσως, ε, απευθείας, είτε εμέσως με περιβαλλοντική διάσταση ή με καταπίεση των πολιτικών ελευθεριών και της ελεύθερης έκφρασης λόγω χάρη στην Κίνα. Ε, το θέμα της ε, Κίνας το θέτω και στην Ολομέλεια από τότε που οι συμπολίτες μας διώχθησαν διότι θεωρήθηκαν αντιφρονούντε από το κινέζικο καθεστώ. Καλό θα ήταν λοιπόν και αυτό να το έχουμε υπόψη μα. Θα υποβάλω λοιπόν πρόεδρε τροπολογίε και θα ήθελε ο συνάδελφο ΕΚ, εφόσον βρισκόμαστε και στην ίδια παράταξη, μπορώ να το πω έτσι, ε, να συνεργαστεί μαζί μα ώστε να ετοιμάσουμε όντω ένα άρτιο κείμενο και να είναι ένα σχέδιο γνωμοδότησης που θα αποσταλεί στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ώστε να πιάσει τόπο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λάινεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ορθό μου φαίνεται και σωστό να συντάξει γνωμοδότηση για την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών για τη σχέση με την Κίνα η δική μας Επιτροπή, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, διότι μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με την Κίνα. Και ευχαριστώ ιδίως ε, τον κύριο Εκ για το σχέδιο γνωμοδοτήσεως, το οποίο νομίζω σημειώνει μερικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Όμως κύριε Φαρία, η Κίνα είναι μεγάλη χώρα. Στην ουσία αποτελείται από πολλές χώρες ένα ενίο σύνολο. Διότι έχει καλές πλευρές που μας αρέσουν και άσχημες πλευρές που δεν μας αρέσουν. Αυτά βεβαίως θα τα περιλάβει στο περιεχόμενο της εκθέσεώς του, της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής, δηλαδή ο κύριος Μπέλτερ. Εν πάση περιπτώσει, ασφαλώς και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι μια σημαντική αξία, βεβαίως και το καθαρό νερό, καθαρό νερό, ο καθαρός αέρας, το καθαρό έδαφος είναι και αυτά ανθρώπινα δικαιώματα. Και φαίνεται πως η κομμουνιστική ηγεσία της μεγάλης αυτής χώρας το έχει κατανοήσει, διότι στο τελευταίο πενταετές πρόγραμμα, από αυτά που ακούσαμε κιόλας από το κομματικό του συνέδριο, κατευθύνονται προς την κατεύθυνση ενός οικολογικού πολιτισμού. Θεωρώ λοιπόν ότι δράτουν, ότι δρούν, συγγνώμη, σωστά, διότι ό,τι συμβαίνει στην Κίνα έχει επιπτώσεις και σε άλλα μέρη του κόσμου και βεβαίως και σε εμάς και ιδίω σε ό,τι αφορά την προστασία του κλίματο και την αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων, βεβαίω έχει άμεση ε, επιρροή αυτό σε εμά, διότι γνωρίζουμε ότι αυτά τα πράγματα είναι ήδη που σπανίζουν και κάθε επιδείνωση από τη χρήση που μπορεί να κάνει η Κίνα σημαίνει μια συνολική επιδείνωση για όλη την ανθρωπότητα. Το ίδιο θα μπορούσε να πει βεβαίως κανείς και για την Ινδία ή και για άλλες μεγάλες χώρες. Αλλά αυτό δεν είναι αντικείμενο της παρούσης η πολιτική κλίματος είναι ένα βασικό τμήμα των προσπαθειών για την διάσωση του κόσμου, των οικοσυστημάτων του κόσμου, ας πω καλύτερα. Οι Κινέζοι εδώ, εξιδίου συμφέροντος κινούμενοι, έχουν κάνει πραγματική μεταβολή, στροφή επιτόπου από μια αμυντική στάση σε μια μάλλον επιθετική στάση. Αυτό είναι καλό. Είναι καλό διότι η τρομακτική ατμοσφαιρική ρήπανση στις κινέζικες πόλεις είναι αυτή η οποία παρεκκίνησε την ε, κομμουνιστική ηγεσία να λάβει μέτρα. Εν τέλει, αυτό μας βρίσκει βεβαίως σύμφωνους. Σε ό,τι αφορά τώρα τις COP, δηλαδή τις ε, διασκέψεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, πρέπει να μιλήσουμε εκεί με καθαρό λόγια με την Κίνα. Στην COP23, ε, στην Βόνη, είδαμε ότι η Κίνα χωρίζει τον κόσμο ολόκληρο ακόμη σε δύο μέρη. Τις βιομηχανικές χώρες που οφείλουν όλες να κάνουν τα πάντα και τις αναπτυσσόμενες χώρες οι οποίες δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα. Και η Κίνα θεωρεί αυτήν ακόμα αναπτυσσόμενη χώρα και όχι βιομηχανική. Νομίζω ότι τουλάχιστον στην COP24 που θα διεξαχθεί στην Πολωνία θα πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα αυτά, θα πρέπει να συμβάλλει η Κίνα και όσο το δυνατόν συντομότερο και θα πρέπει να συμβάλλει και χρηματοδοτικά. Δεν είναι καμιά φτωχή χώρα πλέον η Κίνα, είναι πλούσια χώρα. Και έως τώρα η Κίνα δεν συμμετέχει στο λεγόμενο πράσινο ταμείο. Έχει ιδρύσει ένα δικό της ταμείο. Εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν είναι σωστό. Θα πρέπει να συμβάλλει χρηματοδοτικά στα διάφορα ταμεία που έχουμε ιδρύσει. Η, Κίνα, ε, η Ευρώπη βοήθησε να δημιουργηθεί το σύστημα μείωσης των ε, αερίων θερμοκηπίου στην ε, ε, Κίνα. Ίσως θα πρέπει κάποια στιγμή να συνδεθούν οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας να μπορέσουν, από κάρβουνο δηλαδή, να μπορέσουν να συνδυάσουν τις προσπάθειές τους. Θα μιλήσω και για την κυκλική οικονομία. Η αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων είναι σημαντικό θέμα, αλλά όταν έχετε 1,4 δισεκατομμύρια κατοίκους νομίζω μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα έκλεισε την πόρτα η Κίνα τώρα για τις εισαγωγές ε, αποβλήτων από την Ευρώπη. Το κατανοώ αυτό διότι έχουν και αρκετά σκουπίδια δικά τους. Και εμείς δεν θέλουμε τα δικά, τα δικά μας και τα στέλαμε ως τώρα σε αυτούς. Έχουν λοιπόν δίκιο να το κάνουν. Αλλά τέλος πάντων θα είμαι σύντομος. Ενέργεια και μεταφορές. Τα είπαν αυτά. Η ηλεκτροκίνηση των οχημάτων. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι και μια κίνηση προστατευτισμού, διότι οι μπαταρίες που χρησιμοποιούν τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητά τους δεν επιτρέπεται να προέρχονται από αλλού παρά μόνο από την ίδια την Κίνα. Θα κάνω κάποιες τροπολογίες εν, πάση περιπτώσει για να βοηθήσω να βελτιωθεί το κείμενο του κυρίου Εκ. Ευχαριστώ κύριε Λάινεν και κυρία Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεσή του. Θα παραμείνω στα θέματα που αναφέρονται στο περιβάλλον χωρίς να σημαίνει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα βεβαίως δεν είναι σημαντικά. Αλλά εδώ το θέμα είναι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Και πράγματι εξετάζεται το στρατηγικό θεματολόγιο, οι τομεί συνεργασίας είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, οι ανταλλαγές μεταξύ προσώπων κλπ. Θα ήθελα να καθορίσουμε εμείς το όραμα του μέλλοντος σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μεταξύ Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, να βασίζονται δηλαδή σε μια, σε, μια βάση μεγαλύτερη συνεργασίας. Μου αρέσει το ύφο της εκθέσεως, βρίσκω ότι είναι φιλικό, δεν αξιώνει πράγματα, μιλεί πολύ για συνεργασία και νομίζω ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Νομίζω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε και την άποψη ότι πολύ περισσότερα θα επιτύχουμε αν συνεργαστούμε σε περιβαλλοντικά θέματα αντί να παρεμποδίζουμε ή να επικρίνουμε διαρκώς την Κίνα. Βεβαίω υπάρχουν και τομείς που με ανησυχούν ιδιαίτερω. ω παράδειγμα, επίκαιρο, είναι ζητήματα εναέριων μεταφορών που βλέπουμε η Κίνα να προσπαθεί να υποτιμήσει ορισμένα από τα offset Εκεί νομίζω ότι μπορούμε πράγματι να συνεργαστούμε πολύ στενά σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση του τρόπου χρήσεως των offset. Σε άλλους τομείς της εμπορίας ε, των εκπομπών μπορούμε να κερδίσουμε πολύ περισσότερα πράγματα συνεργαζόμενοι με την Κίνα. Αυτοί έχουν ένα σύστημα το οποίο είναι συμπληρωματικό του δικού μας και μπορούμε έτσι να βαδίσουμε από κοινού προς την κατεύθυνση ενός παγκόσμιου συστήματος αντί να τους κατακρίνουμε διαρκώς διότι δεν τηρούν τη στάση που θα αναμέναμε εμείς από αυτούς. Ε, παραλαμβάνω ότι πολλά περισσότερα θα κερδίσουμε εάν συνεργαστούμε. Χαίρομαι που βλέπω ότι ο εισηγητής καλύπτει κάποια από τα βασικά ε, θέματα. Θα μου επιτρέψει να καταθέσω και εγώ μερικές τροπολογίες και ιδίω ε, σε ό,τι αφορά κανονιστικά συστήματα. Γιατί για μένα εδώ ανοίγεται μια μεγάλη ευκαιρία για τις μελλοντικέ σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών για μια ρυθμιστική σύγκληση. Η Κίνα, όπως έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, έχει δύο επιλογές ή και τρεις αν θέλετε σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση. Είτε θα βάλουν δικά τους πρότυπα, είτε θα ακολουθήσουν το αμερικανικό ε, μοντέλο, είτε το ευρωπαϊκό. Βεβαίως δεν είναι τα ίδια τα πράγματα αυτά, αλλά ε, με τον τρόπο αυτό θα το πράξουν. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ακολουθήσουν το ευρωπαϊκό πρότυπο. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν να τονίσουμε τα πλονεκτήματα που πρέπει να αναμένονται από μια τέτοια κίνηση και να αναπτυχθεί περισσότερο η σύγκληση αυτή. Όταν ρυθμίζουμε τα πράγματα όπως πάμε να κάνουμε τώρα για τα πλαστικά, αυτό θα γίνει αμέσως κατανοητό και θα μπορεί να γίνει και ανταλλαγή με κινέζικα μέτρα, με κινέζικες ρυθμίσεις. Και όπως ορθά αντιλαμβάνεται ο εισηγητής, οι κινέζικες αποφάσεις για τα πλαστικά στην ουσία υπαγορεύουν το τι θα κάνουν και οι υπόλοιποι παίκτες παγκοσμίω. Υπάρχουν και άλλα θέματα όπως η καλή μεταχείριση των ζώων. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα έκθεση στον αγροτικό τύπο του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τον αριθμό εξαγωγών σπέρματος και οαρίων για την γονιμοποίηση ζώων. Οι Κινέζοι θα καταναλώσουν πολύ πολύ περισσότερο κρέας στο μέλλον. Αυτό το είναι για μας και μια ευκαιρία για να μπορέσουμε να τους οδηγήσουμε σε μια σύγκληση και για τις ρυθμίσεις για την ορθή μεταχείριση των ζώων. Θεωρώ λοιπόν ότι η έκθεση έχει καλώς, αλλά θα χρειαστεί κάποιες τροπολογίες. Ευχαριστώ και για την Μάκη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και με τη σειρά μου ευχαριστώ τον κύριο Εκ για την θαυμάσια εργασία που έχει καταθέσει. Παρόλο τον περιορισμό της μιας σελίδας Κατάφερε ωστόσο μέσα σε αυτή τη μία σελίδα να περιλάβει τα πιο σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα που πρέπει να τεθούν επιτάπητος σε συζητήσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Χαίρομαι που βλέπω κάποια πράγματα που γράφει, που τονίζουν την δημόσια υγεία, ιδίως σε ό,τι αφορά την αρθεκτικότητα στα αντιβιωτικά των μικροβίων. Κίνα και Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί είναι υπεύθυνε για μέγα μέρος των ε, αερίων του θερμοκηπίου. Ενίσχυση λοιπόν της συνεργασίας, κοινή ανάπτυξη τεχνογνωσίας είναι πολύ σημαντικά πράγματα και θα προσπαθήσω εγώ να περιλάβω τέτοια πράγματα στι τροπολογίε που θα καταθέσω. Θεωρώ ότι θα πρέπει να αναγνωρίσετε την καλή δουλειά που έχει αρχίσει να κάνει η Κίνα σε πολλούς τομείς αλλά και να την ενθαρρύνεται τη μεγάλη αυτή χώρα να συνεχίσει και με μεγαλύτερη φιλοδοξία. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ορισμένους τομείς συνεργασίας. Αυτή τη στιγμή συνεχίζονται διαπραγματεύσεις για μια συνολική συμφωνία επενδύσεων μεταξύ Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ μάλιστα προτίθεμαι να καταθέσω τροπολογίες για τη συμπερίληψη πολύ ξεκάθαρων διατυπώσεων σε ό,τι αφορά την βιωσιμότητα των επενδύσεων. Και με την νεαρά τράπεζα επενδύσεων και υποδομών ASEAN θα ήθελα για το θέμα αυτό να ζητήσω από τις χώρες μέλη εκείνες που συμμετέχουν στην AIB να υψώσουν τη φωνή τους υπέρ βιώσιμων προτύπων για τις επενδύσεις. Η ανάπτυξη των υποδομών στην Ασία θα απαιτήσει επενδύσεις 3 εκατομμυρίων δολαρίων στα επόμενα χρόνια. Αυτό αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία ή βέβαια και ένα τεράστιο κίνδυνο αναλόγως των πρακτικών που θα επιλεχθούν. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τον σεβασμό μου για την από μακρού διμερή πρωτοβουλία Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας. Χρειαζόμαστε πρότυπα, πρότυπα για την ξυλία και αυτά να επιβληθούν παγκοσμίω. Εδώ Κίνα και Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αποδειχθούν ότι θα είναι ισχυρότατοι σύμμαχοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Άλλος κανείς παρακαλώ που επιθυμεί να λάβει το λόγο. Μήπως κάποιος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλει να απαντήσει. Καλησπέρα σας. Δεν είμαι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά από την ΕΕΔ. Και επειδή αυτό είναι θέμα γενικού ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας, έχω εδώ κάποιους συνάδελφους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μπορούν να με υποστηρίξουν αν χρειαστεί και να με διορθώσουν για πιο συγκεκριμένε απαντήσει αν χρειαστεί. Πάντως, εν γέννη, θα ήθελα να ευχαριστήσω που μας δίνετε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε στην ε, συζήτηση αυτή και να δώσουμε τη δική μας την άποψη για το σχέδιο γνωμοδότησης. Απλώς μια γενική παρατηρήση όπως είπαν και οι προλαλήσαντες. Οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας είναι ποικιλόμορφες. Ε, σφαιρικού χαρακτήρα και καλύπτουν ένα μεγάλο εύρο θεμάτων. Υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία έχουμε κάποια διαφωνία, όμως εν γέννη η συνεργασία μας για, για το περιβάλλον, την ε, ασφάλεια των τροφίμων, την ε, ε, ποιότητα των προϊόντων, εκεί έχουμε ένα θετικό κατάλογο προτεραιοτήτων. Άρα, από αυτήν την έννοια, το σχέδιο γνωμοδότησης αγγίζει κάποια σημαντικά θέματα τα οποία και εμείς θα παρακολουθούμε στην καθημερινή μας ε, συνεργασία με την Κίνα. Πολλά θέματα όπως η συνεργασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχους της για την ανάπτυξη που να είναι απαλλαγμένη από τον άνθρακα, για τη διαχείριση αποβλήτων ή τη συνεισαγωγή αποβλήτων και λιμάτων. Ε, Η γνωμοδότηση αναφέρεται και σε εξελίξεις στην Κίνα ως χώρα. Τα αναγνωρίζουμε και εμείς ως σημαντικά. Οι Κινέζοι πρέπει να κάνουν προσπάθειες για να καλλιεργήσουν τον οικολογικό τους πολιτισμό και τη σχετική νοοτροπία, αλλά η θετική μας στάση προς την, ε, η γενική μας στάση προς την έκθεση αυτή, τη γνωμοδότηση, είναι θετική. Είμαστε θετικά διακείμενοι και ελπίζουμε ότι το τελικό σχέδιο έκθεσης θα αντικατοπτρίζει τον ε, πολύπλοκο χαρακτήρα και το δίκτυο των σχέσεών μας με την Κίνα. Επ' αυτή την έννοια λοιπόν ευχαρίστω να συμβάλλουμε και να συνεργαστούμε μαζί σας για την κατάρτιση της έκθεσης αυτής, αλλά γενικότερα και για όποιο άλλο θέμα άπτεται του περιεχομένου της. Thank Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Εκ. Ευχαριστώ, αγαπητή Πρόεδρε. Έγραψα την γνωμοδότηση υπό το πρίσμα βέβαια των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ασφάλεια τροφίμων, περιβάλλον, δημόσια υγεία. Δεν πήρα δεν στόχευσα στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διότι θεωρώ ότι αυτόν επιλαμβάνονται άλλοι και καλύτερα από μένα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εμείς εδώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος αρχιοθετούμε τα θέματα των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Όμως, η Επιτροπή Περιβάλλοντος θα με τα θέματα περιβάλλοντος. Βέβαια, συνέταξα όντως την έκθεση σε φιλικό τόνο έχω ζήσει έξι χρόνια στην Ασία και τους γνωρίζω καλά τους Ασιώτες, Ασιάτες και θεωρώ ότι διαπραγματεύεται κανείς καλύτερα μαζί τους και έχει καλύτερη επαφή και συνεργασία εάν τους φέρετε φιλικά. Απέναντι στους Κινέζους διόλου δεν να εμφανίζεται κανείς με ένα ρόπαλο στο χέρι και να του χτυπάει στο κεφάλι και μετά να προσπαθεί να επιτύχει ένα καλό αποτέλεσμα. Δεν πρόκειται να επιτύχει. Προσπάθησα λοιπόν να φτιάξω κάτι το οποίο να σας φανεί καλό. Αναμένω με χαρά τις προτάσεις βελτιώσεως που θα υποβάλλετε για να μπορέσουμε τέλει να θέσουμε υπόψη του Κοινοβουλίου ένα σωστό κείμενο. Σας ευχαριστώ πολύ. Η προθεσμία τώρα καταθέσεως τροπολογιών η 6η Μαρτίου στις 11 το πρωί και η ψηφοφορία στις 25 και 26 Απριλίου, 25 ή 26 Απριλίου. Στην ΔΕ Επιτροπή Εξωτερικών προβλέπεται η ψηφοφορία στις 26. έκτου. Το επόμενο θέμα στην ημερησία διάταξη μας, ακολουθεί, μας ε, έρχεται τώρα. Υποδέχομαι τον κύριο Αλέξη Κουστίλ, που είναι διευθυντής του Κέντρου Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, με έδρα τη Λισαβόνα. Πρόκειται για την πρώτη φορά που ακούει η Επιτροπή μας για το κέντρο αυτό συνήθως είναι Επιτροπή Θεμελιωτών Ελευθεριών που ασχολείται με τα θέματα αυτά, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον και για εμάς. Μιλούμε για τις ψυχοτρόπες ουσίες και για το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Υπενθυμίζω ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος έχει καταθέσει πλήρωνες γνωμοδοτήσεις για τι ψυχοτρόπες ε, ουσίες και για τις ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες στη δημόσια υγεία. Υποστηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Επιτροπή και το έργο του παρατηρητηρίου για ε, την αντιμετώπιση των ιών. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ κύριε Γκουστήλ. Μετά από την πρώτη σας παρουσίαση θα έχουμε την ευκαιρία να προβούμε στην ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που με προσκαλείτε εσείς να σας παρουσιάσω ε, κάποιες από τις σημαντικότερες προκλήσεις που έχουν σχέση με τα ναρκωτικά στην Ευρώπη, δεδομένου δε ότι αυτός ο μήνας είναι ο μήνας όπου εδώ και 25 χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την ε, θετική, μάλλον με θετική του γνωμοδότηση ελήφθη απόφαση για την νομοθέτηση και τον κανονισμό που ίδρυσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας. Και πράγματι είναι η πρώτη φορά που ο Διευθυντής του Οργανισμού έχει το ε, προνόμιο να σας παρουσιάσει τις προκλήσεις αυτές. Αντί λοιπόν να σας μιλήσω για το πόσο και, ζωντανός και νέος είναι ο οργανισμό, να μιλήσω περισσότερο για θέματα που ενδιαφέρουν το έργο της Επιτροπής σας. Με δύο λόγια, ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις από τη σκοπιά της ε, δημόσιας υγείας ε, για την Ευρώπη όσον αφορά τα ναρκωτικά. Θα σας τα παρουσιάσω με λίγο περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι η αυξανόμενη διαθεσιμότητα, η καθαρότητα και η, καινοτόμες, ε, η καινοτόμος είσοδος στην αγορά των παράνομων ναρκωτικών που αποτελούν διαμεθοριακό κίνδυνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ε, άλλο πρόβλημα είναι ο αυξανόμενος ρόλος του διαδικτύου και του σκοτεινού δικτύου για τη διάδοση των ναρκωτικών αλλά και όλο και περισσότερο για τις, με τους νέους καινοτόμους τρόπους στον τομέα της πρόληψης και της ε, ε, αντιμετώπισης της χρήσης ναρκωτικών. Κατόπιν έχουμε το αυξανόμενο πρόβλημα των νέων ψυχοδραστικών ουσιών στην Ευρώπη. Ε, πρέπει να σας ε, ενημερώσω ή να σας υπενθυμίσω ότι μέχρι προενός έτους δύο ήταν οι νέες ψυχοδραστικές ουσίες που έμπαιναν στην ευρωπαϊκή αγορά κάθε εβδομάδα. Τις παρακολουθούσαμε από τη Λισαβόνα πάνω από 620 ουσίες ε, σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και είδαμε ότι ε, ο αριθμός ε, αυτών εμφανίζεται όλο και περισσότερο στην ευρωπαϊκή αγορά. Ε, ε, αυτές είναι τα συνθετικά οπιοειδή, η φεντανίλ δηλαδή και άλλες ουσίες, ε, άλλες ομάδες ουσιών που σε κάποια κράτη-μέλη έχουν οδηγήσει σε σημαντικές ή σχετικά σημαντικές αυξήσεις των θανάτων που έχουν σχέση με τα ναρκωτικά. Μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η αλλαγή διεθνώς των πολιτικών σε σχέση με την κάναβη και ένα βασικό πρόβλημα είναι η πατήτηδα ε, γάμα ε, που αφορά τα άτομα που κάνουν ε, ε, που ενέσιμα, χρήση ενέσιμων ναρκωτικών και που μπορούν να προσβληθούν από τον ιό αυτό και που για πρώτη φορά πλέον μπορούν να, να, αντιμετωπιστούν και να θεραπευτούν. Συνεργαζόμαστε με Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ και άλλες γενικές διευθύνσεις και ε, διεθνείς για να ενώσουμε τις δυνάμεις μας να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Εδώ στην περίπτωσή μας αυτή είναι η ομάδα στόχος που βρίσκεται στο επίκεντρο του, ε, του έργου του οργανισμού. Όταν λέω ότι όλο και περισσότερο διατίθενται τα ναρκωτικά στην ευρωπαϊκή αγορά, αξίζει τον κόπο να σας παρουσιάσω τις πρώτες εκτιμήσεις που δημοσιεύσαμε σε συνεργασία με τη Europol πριν από δύο χρόνια. Οι εκτιμήσεις αυτές και ξέρουμε ότι είναι μάλλον χαμηλές. Τουλάχιστον 24 δις ευρώ ε, που είναι το αποτέλεσμα του, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών στην Ευρώπη που βεβαίως ε, ε, ε, χρηματοδοτεί πολλές άλλες δραστηριότητες ε, οργανωμένου εγκλήματος. Το παράδοξο εδώ λοιπόν είναι ότι λόγω των πολλών και αρκετά καλά ανεπτυγμένων τρόπων αντιμετώπισης του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ευρώπη, το παράδοξο είναι ότι είναι πολύ παρόντα τα ναρκωτικά στην Ευρώπη ακόμα. Έχουμε πολλά προβλήματα και πρόβλημα δημόσιας υγείας που σχετίζεται με τη χρήση ναρκωτικών, αλλά ο τρόπος που, έχουν, που χρησιμοποιούνται τα ναρκωτικά έχει αλλάξει πολύ πολύ τα τελευταία 20-25 χρόνια, δηλαδή είναι λιγότερο ορατά, κυρίω σε, συνεργα... σε σύγκριση με το τέλος δεκαετίας του 80 και τον αριθμό των ε, ανθρώπων που πέθαναν από υπερβολική δόση στους δρόμους του κάποιων μεγάλων πόλεων. Μετά οδήγησε αυτό στη δήλωση τη Φραγκφούρτης σε πολλέ καινοτομίε, συμπεριλαμβανομένης και τη θεραπεία και τη αποκατάσταση Ως εκ τούτου τα προβλήματα αυτά δεν είναι πλέον τόσο ορατά. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι δεν υφίστανται. Η εκτίμηση αυτή σα λέει ότι τα ναρκωτικά τελικά εξακολουθούν να υπάρχουν και εξακολουθούν να είναι ε, υπαρκτό πρόβλημα στον τομέα της δημόσιας υγείας. Αν δείτε αυτή την ε, ε, αυτό το, το σχεδιάγραμμα θα δείτε ότι παρατηρήσαμε ότι τα τελευταία τρία χρόνια υπάρχει αύξηση του αριθμού των θανάτων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά και με το πράσινο βλέπετε ότι η αύξηση αυτή ε, έχει γίνει πιο ε, εμφανής σε μεγαλύτερες ηλικίες και αυτό επιβεβαιώνει ότι δεν είναι κάτι ε, μεμονωμένο που αφορά μια ομάδα ηλικίας. Επίσης, η ανταπόκριση ας πούμε, η θεραπεία ε, με οποιοειδή δεν υπάρχουν στοιχεία για την ε, ε, αποτελεσματικότητα και επίσης υπάρχει το πρόβλημα της μείωσης της εκτροπής αυτών των, υποκα... των ουσιών υποκατάστασης και της παράνομης χρήσης αυτών των ουσιών. Ευτυχώς υπάρχουν κάποια αντίδοτα που μπορεί και οφείλουν να χρησιμοποιούνται για την πρόληψη των θανάτων από υπερβολική δόση ανοξών και το ε, νατρολοξών που χρησιμοποιούνται σε 10 κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένων και σε κάποιες περιπτώσεις είναι, ε, ε, είναι διαθέσιμα για τις υπηρεσίες δίωξης που αντιμετωπίζουν ή διαλύουν κάποια εργαστήρια όπου θα μπορούσε η έκθεση σε κάποια συνθετικά οπιοειδή να θέσει εκείνο τη ζωή τους. Υπάρχουν 7 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 8 αν συμπεριλάβουμε και την Ελβετία τη ευρύτερη, της ευρύτερης Ευρώπης που δημιούργησαν ε, ε, αίθουσα επιτηρούμενης χρήσης ναρκωτικών σε συνεργασία με άλλα προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αξιολογείται η προσπάθεια, συντάσσεται ένα έγγραφο για να θεσπιστούν ε, τα κριτήρια και οι βέλτιστες πρακτικές. Αυτές είναι κάποιες από τις απαντήσεις που σήμερα έχουν ε, αναπτυχθεί και μελετώνται. Αξίζει τον κόπο να επισημάνουμε ότι προς το παρόν τουλάχιστον και εδώ αυτό συνεισφέρει στο παράδοξο που ανέφερα προηγουμένως ότι η χρήση ναρκωτικών δεν είναι τόσο εμφανής όσο στο παρελθόν. Έχουμε 630.000 ανθρώπους που παίρνουν θεραπεία υποκατάσταση ναρκωτικών στην Ευρώπη. Σε αρχές δεκαετίας του 90 ο αριθμός τους ήταν ούτε καν 20.000 αυτοί. Τελείωσε ο χρόνος μου διαπιστώνω, λέει ο μιλητής. Έχουμε επίσης τη σύγκριση 20.000 με 630.000. Έχουμε άτομα που παρακολουθούν και άλλους τρόπους θεραπείας. Τώρα η μείωση των κρουσμάτων HIV συνεχίζει να ε, συνεχίζει, τουλάχιστον όσο σε σχέση με αυτούς οι οποίοι παίρνουν ενέσιμα ναρκωτικά. Έχουμε φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο της δεκαετίας. Εν μέρη αυτό οφείλεται στις ε, παρεμβάσεις για τη μείωση της βλάβης και για τις διάφορες δοκιμές, ε, για τα τεστ που υπάρχουν στους χρήστες ναρκωτικών. Σκοπός μας είναι να, να συνεχίσουμε και να αναπτύξουμε την περαιτέρω τη διαθεσιμότητα θεραπείων Επίσης αναφέρθηκα στην, ε, στον επιπολασμό της υπατήτηδας. Θα δείτε ότι υπάρχει τεράστια διακύμανση στην Ευρώπη ε, σε σχέση με τον αριθμό των χρηστών ναρκωτικών που είναι θετική σε υπατήτηδα Γ από 16 έως 84 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι και εδώ όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις δεν υπάρχει μία μοναδική προσέγγιση και χρειαζόμαστε τεκμήρια για να στηρίξουμε το σχεδιασμό εθνικών πολιτικών και παρεμβάσεων. Ανέφερα και δεν θα επισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά εισαγωγικά όταν αναφέρθηκα στα βασικά σημεία και τις βασικές προκλήσεις έχουμε αυξανόμενη διαθεσιμότητα ναρκωτικών στην Ευρώπη. Αυτό ισχύει για την κοκαίνη τόσο όσον αφορά την ποσότητα αλλά και την καθαρότητά της. Επίσης ισχύει ε, και παρατηρείται αυτό μέσω των, της επιδημιολογίας των λιμάτων σε κάποιες πόλεις υπάρχει μεγάλες, υπάρχουν μεγάλες συγκεντρώσεις υπολοιμάτων κοκαίνης. Το ίδιο ισχύει και για το έκσταση και θα ήταν ε, ενδιαφέρον ίσως για σας να μάθετε ότι το έκσταση είναι περισσότερο διαθέσιμο και σε ψηλότερες συγκεντρώσεις από, από τις πριν από 10 χρόνια και αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι η παραγωγή του έκσταση βρήκαν τρόπο να βρουν νέους, νέες πρόδρομες ε, χημικές ουσίες για να αποφύγουν ε, την προσπάθεια της δίωξης να αντιμετωπίσουν τους, τις πρόδρομες ουσίες. Παραδείγματος χάρη, πριν από 15 χρόνια το, ε, ο οργανισμός ξεκίνησε μια προσπάθεια γιατί είχε βρεθεί χάπια έκσταση σε ένα φεστιβάλ ροκ στο Βέλγιο με 65 μιλιγκράμμ ουσίας. Τώρα βρίσκουμε μέχρι 180 μιλιγκράμμ ε, στα ε, χάπια. Βλέπετε λοιπόν ότι η κίνδυνη για την υγεία είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στο παρελθόν. Και για να ολοκληρώσω θα ήθελα να επισημάνω ένα από, μία από τις βασικές προκλήσεις που εξελίσσονται μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα στην Ευρώπη είναι οι παγκόσμιες πολιτικές σε σχέση με την κάναβη. Ε, στην Αμερικανική Ήπειρο γίνονται σημαντικές αλλαγές. Στην Ευρώπη υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στη χρήση και στην ε, ρύθμιση της χρήσης της κάναβης. Πολύ διαφορετική από τις ΗΠΑ. Δεν υπάρχει κυβέρνηση που να στηρίζει προς το παρόν την πλήρη νομιμοποίηση και οι εξελίξεις και οι πρόσφατες ε, ε, εξελίξεις έχουν δείξει ότι πρέπει να παρακολουθούνται οι επιπτώσεις σοβαρά. Και ξέρω επίσης ότι σήμερα θα συζητηθεί και το άλλο θέμα, το θέμα των ε, φαρμάκων με βάση την κάναβη. Συνήθως μιλάνε για ιατρική, κάναβη για ε, θεραπευτικούς σκοπούς, αλλά υπό με θεραπευτικούς ή ιατρικούς όρους θα ήταν καλύτερο να μιλάμε για φάρμακα με βάση την κάναβη και όπως σε όλα τα θέματα έτσι και εδώ υπάρχει μεγάλη διαφορά στην κατάσταση και στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ό,τι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά με δύο λόγια ήθελα να σας πω η εξέλιξη, η πιθανή εξέλιξη των θανάτων από ναρκωτικά, κυρίως που ε, έχουν σχέση με την ομάδα των φενταλινών, είναι πολύ σημαντική. Μια εικόνα για σας. Το 2016 στην Ευρώπη ε, έγιναν υπήρχαν 8.000 θάνατοι από υπερβολική δόση. Ηνωμένε ΗΠΑ το 2016 ήταν 66.000 ε, αυτοί οι οποίοι πέθαναν από υπερβολική δόση ε, οπιοειδών και τώρα οι πρόσφατε πληροφορίε που έλαβα από του συναδέλφου από τις ΗΠΑ πριν από μια εβδομάδα όταν συναντήθηκα με το Εθνικό Ινστιτούτο κατάχρηση Ναρκωτικών είναι 170.000 θάνατοι από υπερβολική χρήση ε, οπιοειδών την ημέρα είμαστε σε καλύτερη θέση από ότι στην Ευρώπη. Βεβαίως, σημαίνει αυτό ότι ποτέ δεν θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάποιες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν εκεί. Τουλάχιστον τα δεδομένα που παίρνουμε από το ε, σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης των νέων ψυχοδραστικών ε, ουσιών δείχνει ότι τα φεντανίλ έρχονται στην Ευρώπη από τις 32 φεντανίλε που ελέγχονται ε, στην Ευρώπη από το 1997 έχουμε περίπου 25 στην αγορά τα τελευταία δύο χρόνια. Βρέθηκαν 25 στην αγορά τα τελευταία δύο χρόνια. Οι κίνδυνοι υπάρχουν, οι προκλήσεις υφίστανται και η σημασία της συγκέντρωσης και οικοδόμησης των τεκμηρίων για την πολιτική ε, ε, είναι εξίσου σημαντική και τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρουσίαση κύριε Διευθυντά. Ε, υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θέλει το λόγο. Η κυρία Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστούμε για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Θα ήθελα να σας ε, θυμίσω την πρώτη διαφάνεια που μας δείξατε. Έναν από τους τομείς, τα παιδεία που αναφέρατε εκεί, ήταν η επιρροή του διαδικτύου και του σκοτεινού διαδικτύου και αναφέρατε ότι η χρήση ναρκωτικών δεν είναι τόσο εμφανής στο παρελθόν. Αλλά σαφώς εδώ το ίντερνετ και το darknet παίζουν σοβαρό ρόλο. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι ο ρόλο του σκοτεινού διαδικτύου, του αδιαφανούς διαδικτύου, ιδίω ό,τι αφορά του νέου φοιτητέ σε διαφορετικέ χώρε και βεβαίω και στα κράτη-μέλη μα. Καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν ευθυνότερα προϊόντα που μπορούν να αγοράσουν, ανώνυμα μάλιστα, από απόσταση, οπότε ναι, το Darknet παίζει έναν σοβαρότατο ρόλο στην παράνομη πώληση ναρκωτικών και δυστυχώς βλέπω ότι σε μεγάλο ρυθμό κρατών μελών δεν αντιμετωπίζεται το θέμα απευθείας όπως θα έπρεπε. Από την δική σας λοιπόν την εμπειρία και από τους τομείς που αναφέρατε. Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες από αυτού. Τι τάσεις γνωρίζετε ότι υπάρχουν. Τι παρατηρείτε. Ποιε είναι οι υποθέσει που περισσότερο σα ανησυχούν, Είστε ικανοποιημένο με τον τρόπο που τα κράτη-μέλη μα και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του ε, διαδικτύου και του σκοτεινού διαδικτύου. Μπορείτε να μας δώσετε πληροφορία, πληροφορίες για ουσίες που αγοράζονται στο διαδίκτυο και που δεν είναι απαραίτητο παράνομες αυτές καθεαυτές αλλά έχουν παρόμοια αποτελέσματα και επιπτώσεις με τα παράνομα, με τις παράνομες ναρκωτικές ουσίες. Θέλετε να απαντήσετε στις δύο ερωτήσεις τώρα ή μετά, αφού ακούσουμε κι άλλες. Να απαντήσω καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ντάλη για τις ερωτήσεις σας και τα σχόλιά σας. Έχω κάποια πράγματα να σας αναφέρω τώρα και μπορώ και να σας στείλω λεπτομέρειες γραπτός, δεν τα ξέρω απ' έξω. Ε, πέρσι δημοσιεύσαμε δύο σημαντικές εκθέσεις για το Darknet. Έχετε δίκιο, το διαδίκτυο παίζει πολύ σοβαρό ρόλο, όχι μόνο στις πωλήσει και την διακίνηση των ίδιων των ναρκωτικών, αλλά κυρίως στις παράνομες ουσίες και σε αυτές που είναι ακόμη ε, νόμιμες, δεν έχουν απαγορευτεί. Υπ' αυτήν την έννοια, και επειδή προηγουμένως μιλούσατε για την Κίνα, από τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, σε συνεργασία με την Ευρωπόλ, και αυτό επιβεβαιώνεται και από τις ΗΠΑ και τις πληροφορίες τους, οι περισσότερες αμφεταμίνες έρχονται από την Κίνα. Μερικέ μόνο από την Ινδία, αλλά οι περισσότερε αμφεταμίνε είναι κινέζικης προέλευση. Μεγάλη πρόκληση λοιπόν για τι διοικητικέ αρχές είναι ότι στο λιμάνι του Ρότερνταμ έχουμε 20.000 ε, εμπορευματοκιβώτια καθημερινά σε κίνηση. Ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσει κανείς σοβαρά αυτό το πρόβλημα είναι με καλύτερες μυστικές πληροφορίες, διότι μόνο τα τεχνικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας δεν επιτρέπουν να σκανάρουμε το καθένα από αυτά τα κοντέινερ, από τα εμπορευματικά Οπότε αυτό είναι ένα πρόβλημα ήδη. Η πρώτη έκθεση που το κέντρο μας δημοσίευσε για την αγορά ναρκωτικών στο ίντερνετ το 2016 λέει βάσει της ανάλυσης που κάναμε την Απροπόλ και κάποιους εμπειρογνώμονες ότι προς στιγμήν αλλά ξέρετε ότι η αγορά αυτή διαρκώς μεταλλάσσεται. Προ στιγμή, το μεγαλύτερο μέρος των κεντρικών μέσω διαδικτύου σχετίζεται με τοπικέ αγορέ, μικρέ ποσότητε, δηλαδή και εμπόριο που χρησιμοποιεί και το γεωγραφικό εντοπισμό με εφαρμογές, apps, που επιτρέπεται η διοργάνωση των πωλήσεων και μάλιστα με τρόπο ιδιαίτερα προηγμένο. Αυτά αναπτύσσονται όμω πιο πολύ σε τοπικό επίπεδο, σε μικρή ακτίνα και κατά πάσα πιθανότητα όχι σε όλε τι ευρωπαϊκέ πόλει. Ακόμη και σε μεγάλε ευρωπαϊκέ πόλει τα πάντα εξαρτώνται από τη χρήση του διαδικτύου. Κατά πόσον δηλαδή χρησιμοποιείται το ίντερνετ ευρέω σε αυτέ τι πόλει. Αυτό ήταν το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουν ό,τι μπορούν για να καταπολεμήσουν το φαινόμενο, αλλά από τη δική μας την οπτική γωνία και αυτό εν μέρη είναι κάτι που γίνεται και σε εθνικό επίπεδο, η δημιουργία του ειδικού κέντρου για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος στην Europol είναι, στην Ευρωπόλη είναι πολύ σημαντικό. Ε, το εγκλήμα δεν είναι σημαντικό μόνο για τη διακίνηση των ναρκωτικών και τα παράνομα ναρκωτικά, αλλά για να ενισχύσουμε όλε τι δυνατότητέ μα στην Ευρώπη. Στην πιο πρόσφατη εκθεσή μα που δημοσίευσαμε πέρσι, αυτό που λέμε από κοινό με την Ευρωπόλη είναι ότι αυτή η μεγαλύτερη η στήριξη των δυνατοτήτων μα, σε συνεργασία με τι διαδικτυακέ αρχέ, για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του διαδικτύου και του κυβερνοεγκλήματο, ε, μα φέρνει στα πορίσματα τη έκθεση για τον Darknet, για το σκοτεινό διαδίκτυο, που δημοσιεύτηκε πέρσι τον Νοέμβριο. Και που για πρώτη φορά κάνει μια συνολική αποτίμηση αξιολόγηση των ε, προεκτάσεων που έχει το σκοτεινό διαδίκτυο, όσων γνωρίζουμε τουλάχιστον και έχουμε καταφέρει να συλλάβουμε, να σταματήσουμε. Και αυτά έχουν πολύ σημαντικά μεγάλη σημασία όχι μόνο για τα κάτι μέλη σε εθνικό επίπεδο, αλλά και για τι διοκτικέ αρχέ. Πρέπει να ενισχύσουμε τι δυνατότητε προστασία μα. Και αυτό συμπεριλαμβάνει βεβαίω την προστασία από τη διακίνηση ναρκωτικών. Για να ολοκληρώσω αυτή τη σύντομη απάντηση. Να, να ξαναπώ ότι μόλι επιστρέψω στη Λισαβόνα θα σα στείλω και περισσότερε λεπτομέρειε. Απλώ δύο πολύ σύντομε διευκρινήσει. Πρώτον, το διαδίκτυο μπορεί να είναι ένα εργαλείο για τα πάντα στην ουσία. Δηλαδή μπορεί να φέρει το καλύτερο ή το χειρότερο. Όλο και περισσότερο μάλιστα χρησιμοποιείται για να στοχεύσουμε τους νέους για προγράμματα πρόληψης. Σε κάποια προγράμματα Λόγω χάρη στην Γερμανία υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα. Σε κάποιε χώρε γίνονται γνωστέ κάποιε θεραπείε αποτοξίνωση. Ή για κάποιου που δεν θέλουν αυτόν χρήστη ουσιών, για την ενέσιμη ε, ηρωίνη, για το τι είναι τζάνκι ας πούμε, αυτό είναι ε, κάτι που μπορεί μέσω του διαδικτύου να τους ευαισθητοποιήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και μάλιστα μπορούμε να εντοπίσουμε και τις βέλτιστες πρακτικές μέσω του διαδικτύου. Και τελευταία μου παρατηρήσε για το όλο σας ερώτημα και ισχύει για όλα αυτά που είπα. Το πρώτο πρόβλημα στην Ευρώπη σε αυτόν τον τομέα, όπως και στη ΣΥΠΑ, είναι η υλοποίηση. Έχουμε πολλή γνώση για τις βέλτιστες πρακτικές. Δεν τα ξέρουμε όλα, σίγουρα. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά ακόμα και απορίες. Όμως, βάσει των όσων διαθέτουμε, μπορεί, θα μπορούσε και θα έπρεπε να γίνει καλύτερο σχεδιασμό ε, τη στατικική που θα χρησιμοποιούμε, τη παρέμβασή μα. Και αυτό είναι μια από τι προτεραιότητε του οργανισμού μα ε, ε, για την ερχόμενη τριετία σε συνεργασία και με την DG Center. Ευχαριστούμε ο κύριος Φλάναγκα. Ευχαριστώ. με ενδιαφέραν πάρα πολύ αυτά που είπατε Δεδομένου του τίτλου, του ονόματος του οργανισμού σας, υποθέτω ότι το ενόπνευμα και η κατάχρηση ενόπνευματος ε, που είναι αυτός που σκοτώνει κυρίως τον κόσμο σας ενδιαφέρει. Υπάρχει αυτό το 24 δισεκατομμύρια σε σχέση με την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών στην Ευρώπη. Αλλά ε, εγώ ξέρω ότι 400 δισεκατομμύρια έχουν σχέση με το αλκοόλ και βεβαίως έχουν σχέση με ε, ε, ε, πάσης είδεως ίσης βίας, όπως επίσης και διάλυση οικογενειών. Γιατί αυτά δεν τα περιλαμβάνετε στα διαγράμματά σας. Δεν θεωρείτε η εξάρτηση αυτή βλαβερή ανάλογα με το λόγο του, βλαβερού, του νομικού τους καθεστώτος. Ποια είναι η γνώμη σας για το αλκοόλ. Δεν ξέρω αν υπήρχαν νέοι που θα άκουγαν ε, εδώ αυτή την, παρα... την παρουσίαση θα έλεγαν γιατί δεν υπάρχει το αλκοόλ σε αυτά που λέτε. Επίσης, ε, θα με ενδιαφέρε να ακούσω την άποψή σας για την ε, επιτυχία της ανάκλησης της απαγόρευσης στις ΗΠΑ όσον αφορά την κάναβη και κυρίως το θέμα της φορολόγησης που ε, πηγαίνει τώρα στα εκπαιδευτικά συστήματα, στα σχολεία, στην καθαρότητα του προϊόντος. Τώρα ο κόσμος ξέρει τι χρησιμοποιεί. Το γεγονός ότι δεν έχει προσμίξεις από μια σειρά από ε, ε, χημικές ουσίες, όπως επίσης δεν έχει μουχλά ε, μείωση ε, ως εκ τούτου των ναρκωτικών και μείωση του, ε, του αριθμού των ανθρώπων οι οποίοι οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ και γενικά έχει μειωθεί ο αριθμός των, των χρηστών ναρκωτικών. Αυτές είναι βασικές, βασικές επιτυχίες όσον αφορά τα βασικά δεδομένα, τις βασικές πληροφορίες. Διαρωτώ με, τι είδους πληροφορίες θα χρειαστούμε για να σταματήσουμε σταματήσουν αυτά. Ή οι πληροφορίες είναι απάντηση. Εγώ κάνω εκστρατεία και, έχω στην Ιρλανδία προβάλλει ένα... Ε, νομοσχέδιο για την νομοποίηση της κάναβης έχω δύο φορές φυλακιστεί και στις δύο φορές ε, Κανείς ε, ε, μιλήσατε για σωστές πληροφορίες. Εμένα ε, πριν με βάλουν στο κελί ε, με έψαξαν, ε, ε, με γύμνωσαν, με έψαξαν με στις σωματικές μου κοιλώτες παντού. Με πέταξαν στο κυλί και το μόνο που έκανα μαζί με τον άνθρωπο που ήταν εκεί, καπνίσαμε ένα τσιγάρο. Λοιπόν, πώς ε, περιμένετε να κερδίσετε την υπόθεση αυτή μέσω της συγκέντρωσης πληροφοριών. Μήπως θα πρέπει να σταματήσουμε να βαράμε το κεφάλι μας στον τοίχο γιατί δεν θα ε, γκρεμιστεί ο τείχος αλλά εμείς θα πάθουμε πονοκέφαλο. Πολύ θα με ενδιαφέρει να ακούσω τι έχετε να πείτε επί όλων αυτών. Ευχαριστούμε κύριε Φλάναγκαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Φλάναγκαν. Πολλές οι ερωτήσεις σας, οπότε θα προσπαθήσω να τις θέσω με τη σειρά, να απαντήσω με τη σειρά που τις θέσατε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το αλκοόλ είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, ναρκωτικό κατάχρησης, γιατί δεν αναφέρεται στα σχεδιαγράμματα και στις εκ, εκθέσεις του οργανισμού μας. Συμπεριλαμβάνεται σε κάποιες από τις εκθέσεις όταν μιλάμε για την πολλαπλή χρήση ε, ουσιών, ε, ε, συνδυασμός αλκοόλ και ναρκωτικών. Πολύ συνήθι στην περίπτωση της χρήσης κάναβης, αλλά όχι αποκλειστικά, γιατί δεν μιλάμε περισσότερο. Φοβάμαι λόγω του ότι δεν έχουμε την εντολή να το κάνουμε. Δεν σημαίνει ότι δεν μας ενδιαφέρει καθόλου το θέμα. Όπως γνωρίζετε όλοι πρέπει να ε, ε, παραμείνουμε εντός των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών μας. Παρά τα αυτά, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ σημαντικό θέμα. Η, πολυ... πολλαπλή χρήση ναρκωτικών είναι σημαντική από πολλές απόψεις. Επιπλέον, φέτος η Κομισιόν προετοιμάζει την εξωτερική ε, αξιολόγηση του Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, επειδή θα είναι τα 25 χρόνια, και θα γίνει η αξιολόγηση και μετά τη δημοσίευση των ε, συμπερασμάτων και συστάσεων από πλευράς ε, της Επιτροπής θα γίνει ανάλυση και αξιολόγηση αν και κατά πόσον θα πρέπει να τροποποιηθεί η εντολή του, ε, του κέντρου παρακολούθησης και να συμπεριλάβει το αλκοόλ και άλλες ουσίες και εδώ σας καλώ να εκφράσετε την άποψή σας όσο το δυνατόν πιο έντονα. Ξέρω ότι ο συνάδελφος Κομισιόν θα μιλήσει μετά από μένα μπορεί να σας στείλει ή μπορείτε εσείς να τη στείλετε στείλετε στοιχεία. Πιστεύω ότι τα μέλη της Επιτροπής έτσι και αλλιώ θα κληθούν να απαντήσουν στο ερώτημα σε σχέση με την έρευνα των αξιολογητών. Σας παρακαλώ λοιπόν να εκφράσετε την υποστήριξή σας. Δεν είναι προσπάθεια να αποφύγουμε το θέμα επί της ουσίας δεν μου επιτρέπεται να ασχοληθώ περισσότερο, να επενδύσω περισσότερο αποκλειστικά για το αλκοόλ. Το καλύπτουμε και το λαμβάνουμε υπόψη μας, αυτό είναι σίγουρο. Το τελευταίο θέμα, επίσης σημαντικό, γιατί όλες οι επιτροπές ε, ε, κοιτάνε προς το προϋπολογισμό και των διαφόρων οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς εργαζόμαστε ιδιαίτερα για το συγκεκριμένο θέμα των σχολείων, την, έκθεση, την έρευνα ESPAT, που είναι κομμάτι των δραστηριοτήτων που ζήτησαν από τον οργανισμό μας τα κράτη-μέλη και το θέμα της χρήσης αλκοόλ μεταξύ των νέων ηλικίας 15 και 16 ετών καλύπτεται. Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες, θα σας στείλω την έκθεση μόλις επιστρέψω στη Λισαβόνα την ερχόμενη εβδομάδα, θα σας στείλω την τελευταία έκθεση που ε, δημοσιεύσαμε πέρσι, θα δείτε ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία. Το θέμα είναι πώς θα χρησιμοποιηθεί. Περνάω στο δεύτερο θέμα των σχολείων και των ερωτήσεών σας που αφορά τις επιπτώσεις της νομιμοποίησης της κάναβης για ψυχαγωγική χρήση σε κάποιες ε, πολιτείες των ΗΠΑ. Επιστρέφω από μία αποστολή εκεί την περασμένη εβδομάδα. Είχα κάποιες συναντήσεις στη Ουάσιγκτον με κάποιους συναδέλφους, συμπεριλαμβανομένου και του Εθνικού Ινστιτούτου Κατάχρησης Ναρκωτικών. Επισκέφθηκα τα προγράμματα και έκανα συναντήσεις στο Ντένβερ του Κολοράντο. Αυτό που μπορώ να σας πω επ' αυτού είναι πρώτον, εξακολουθώ υπάρχουν λίγα δεδομένα και λίγες εκθέσεις που επιτρέπουν ουσιαστική αξιολόγηση της επιτυχίας ή μη ή εν πάση περιπτώσει των επιπτώσεων γιατί στις περιπτώσεις αυτές μιλάμε για δημόσια πολιτική και άρα οι επιπτώσεις δεν είναι πάντα λευκές, άσπρες ή μαύρες, υπάρχουν και κάποιες ενδιάμεσες καταστάσεις. Αυτό που είναι ενδιαφέρον και δυστυχώς δεν υπάρχουν ε, συγκριτικά κριτήρια ακόμα. Στις Ηνωμένε Πολιτείε δεν υπάρχει μία πολιτεία ή ακόμα και στην Ουρουάη που να έχουν προετοιμάσει τα συγκριτικά στοιχεία, να έχουν κάνει στατιστικές μελέτες και έρευνες πριν την αλλαγή της νομοθεσίας. Αυτό που σημαίνει ότι είναι δύσκολο να γίνουν συγκρίσεις και είναι λίγο επικίνδυνο το θέμα. Πρέπει λοιπόν να τα παίρνουμε με, ε, ε, με λίγο με προσοχή. Σε κάποιες ομάδες ηλικιών η αύξηση έχει αυξηθεί η χρήση των ναρκωτικών, ας πούμε στο Κολοράντο. Ε, μοιάζει ότι σε αλλού ότι δεν έχει αυξηθεί αλλά δεν έχει μειωθεί λόγω της ε, νέας νομοθεσίας. Είναι στην ομάδα των νέων κάτω των 18 ετών. Αλλά αν μιλήσετε με αυτούς που είναι υπεύθυνοι, ας πούμε, οι υπεύθυνοι του ιατρικού τομέα θα, δει, θα σας πούν ότι η αύξηση συνέβη νωρίτερα όταν ε, λήφθη απόφαση για την θεραπευτική κάναβη, γιατί η θεραπευτική κάναβη στο Κολοράντο δεν ήταν και τόσο θεραπευτική. Και αν δείτε και τα νούμερα για το πόσοι επετράπησαν επιτράπει να ε, πάνε να πάρουν ε, κάναβη για ιατρική χρήση, τα νούμερα αυξάνονται πάρα πολύ. Άρα, αν έχει υπάρξει επίπτωση στη χρήση των ναρκωτικών μεταξύ των νέων, αυτό μάλλον προκλήθηκε από την νομοθετική αλλαγή που αφορά την ιατρική χρήση της κάναβης και αυτό είναι, έχει σχέση με την Ευρώπη γιατί Εκεί δεν έγινε πραγματικά για ιατρικούς σκοπούς και δεν επιβλήθηκε με σοβαρότητα. Το γεγονός ότι μέχρι τούδες αυτή την ομάδα ε, ηλικίας δεν έχει αυξηθεί σημαντικά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ε, ληφθούν μακροχρόνια συμπεράσματα. Ε, θα επανέλθω αν θέλετε, αλλά δεν θέλω να σας καθυστερήσω περισσότερο. Ε, εν πάση αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι όταν πας εκεί, ό,τι και αν είναι η άποψή σου και ο σκοπός της ε, ε, επίσκεψης, έχουμε και μια, μια νέα έκδοση που προετοιμάζουμε φέτος για την ιατρική ε, κάναβη. Εμείς ως οργανισμός πρέπει να βοηθούμε όλους τους, αυτούς οι οποίοι λαμβάνουν αποφάσεις, ευρωπαίους, ευρωπαϊκούς οργανισμούς ή εθνικούς οργανισμούς με τεκμήρια, με στοιχεία, με τεκμηρίωση σε αυτού λείπει. Διαβάζει κανείς ε, για την κάναβη και λέει ας πούμε ότι τώρα όποιος παίρνει κάναβη μπορεί να περπατάει πάνω στο νερό όπως ο Ιησούς. Όχι, πρέπει να ληφθούν, ε, να δοθούν τεκμήρια, τεκμηριωμένες, ε, ε, τεκμηριωμένα στοιχεία. Αλλά ε, οι αποφάσεις είναι πολιτικές. Πρέπει όμως να ε, δίνονται ε, επιστημονικά δεδομένα που θα βοηθήσουν. Δεν έχουμε αποδεικτικά στοιχεία που να λένε προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Εγώ αυτό που το οποίο πιστεύω ότι φοβίζει, ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες δεν ξέρουν τι θα πάθουν. Είναι νέες επικίνδυνες συμπεριφορές λόγω των νέων προϊόντων και τις νέες κάψουλες παραδείγματος χάρη που χρησιμοποιούνται ε, που έχουν 65 έως 95% συγκέντρωση TLC. Αν έχει σε αυτό το υγρό που μπαίνει ε, για το vaping ας πούμε ή δεν προβλέπεται από η χρήση αυτή από τους νομοθέτες και αυτό ενδεχομένως μπορεί να, να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία. Οι Αμερικανοί είναι πολύ ρεαλιστές και πιστεύω ότι αυτά θα τα αντιμετωπίσουν και θα προσπαθήσουν να τα προλάβουν. Αλλά προς το παρόν αυτό ανήκει στη νέα κατηγορία των νέων κινδύνων για την υγεία και ε, επειδή ήταν, ε, δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν πρέπει να αντιμετωπιστούν και το ίδιο περίπου ισχύει με τα βρόσιμα. Σημείωσα τις ερώτησή σας. Αν ξέχασα κάτι, υπόσχομαι ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα σας στείλω ένα mail με την, ε, με την έκθεση. Ευχαριστώ. Thank you very much. Uh, it's great. Ευχαριστώ πολύ. Uh, because it's really very interesting and I'm sorry that we did not have to... Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Σήμερα έχω ε, μάθει πολλά πράγματα από τις ε, συζητήσεις μας σας. Θα έρθω κυρίως στα SDG και στην υπατήτητα. Το Ευρωκοινοβούλιο με επιτυχία έχει εγκρίνει ψηφίσματα σχετικά με τις ασθένειες αυτές, τις οποίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει τη σημασία που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί την, ε, την πρόοδο των ε, βιώσιμων στόχων για την καταπολέμηση της υπατήτητας και την επάρκεια των ε, δεδομένων παρακολούθησης στι διάφορε χώρε μέλη. Είναι ενθαρρυντικό που βλέπουμε σύμφωνα με την ανταπόκριση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων οργάνων αποδίδει για την δημιουργία ενός συνόλου δικτών που θα επιτρέπουν την επίτευξη των στόχων για την ε, υπατητήδα και άλλες σχετικές νόσους μέχρι το 2030. Λόγω της απουσίας ή όπως είπα πριν της ανεπάρκειας των δεδομένων για την ιώδη υπατήτηδα στις χώρες μέλη, σε ποιο βαθμό το κέντρο EMCDDA αναμένει οι δείκτες αυτοί να βελτιώσουν την ποιότητα των διαθεσίμων δεδομένων για την ιώδη υπατήτηδα και για την φυματίωση. Κατά πόσον θεωρείτε ότι είναι πιθανόν οι χώρες μέλη να χρησιμοποιήσουν πράγματι τους δείκτες αυτούς για να παρακολουθήσουν επιδημολογικά την υπατήτηδα και όλες τις διαδοχικές φάσεις της παροχής φροντίδας. Ε, γνωρίζω ότι δεν μπορείτε να προβλέψετε το μέλλον, αλλά ποια είναι η προσωπική σας άποψη για τους νέους αυτούς δείκτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Βάχ. Πολύ σημαντικό θέμα αυτό που αναφέρετε και ιδιαίτερα αγαπητό σε μένα, διότι έχω ε, συνεργαστεί με ανθρώπους που έχουν υπατήτηδα ή που ε, ε, την έχουν δυστυχώς αποκτήσει από τη χρήση ναρκωτικών και όταν μιλώ με συναδέλφους μου των χωρών μελών εκπλήσωμαι και μια φορά βλέποντας ότι σε ορισμένα από τα κέντρα θεραπείας αντιμετωπίζουν λίγο πολύ τις ίδιες δυσχερίες όπως και προ 15-20 ετών. Δηλαδή τελικώς ποιοι είναι οι παράγοντες, τι συμβαίνει. Και αυτό είναι από τα ερωτήματα τα οποία θα θέσουμε στους εαυτούς μας αλλά και στις χώρες μέλη για τα επόμενα δύο χρόνια. Έχουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα για την στήριξη των δράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του EFCDC για την ε, συμβολή στην επίτευξη των στόχων της χιλιετίας. Τι μπορώ να πω για τους δείκτες. Το θέμα είναι δύσκολο, διότι σήμερα, λόγω και της μεγάλης οικονομικής κρίσης του 2008 και των δυσμενών συνεπειών της στους δημόσιους προϋπολογισμούς και ιδίως προϋπολογισμούς για την υγεία των χώρων μελών. Δεν είμαι βέβαιος ότι οποιοδήποτε ευρωπαϊκό όργανο μπορεί να μιλήσει τώρα στις χώρες μέλη για να τους πει «Κοιτάξτε, θέλουμε πιο πολλά χρήματα για πιο πολλούς δείκτες». Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και για να είμαι και ειλικρινής, ε, εδώ δεν ασκώ καμιά κριτική στις χώρες μέλη ή σε κανέναν άλλο. Υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εθνικοί προπολογισμοί πολλών χωρών μελών και ασφαλώς το αποτέλεσμα αυτού είναι ότι ένας από τους τρόπους για να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό είναι πρώτα να διασφαλιστεί ότι θα αποφύγουμε την επικάλυψη μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων και άλλων διεθνών οργανισμών. Και γι' αυτό θεωρώ πολύ σημαντική εξέλιξη την στενή συνεργασία μεταξύ ESCDC, EMCDDA CDDA και την Γενική Διεύθυνση Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το EMCDDA όπως και η Επιτροπή σας δεν συνδέονται τόσο στενά με την ε, Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ, αλλά επειδή έχω διοριστεί, ε, μάλλον από τότε που διορίστηκα ε, ε, Διευθυντή έχω αυξήσει τη συνεργασία και με την Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ και με την δική σα επιτροπή και πολύ χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να συνεργάζομαι μαζί σας. Βέβαια δεν μπορώ να προβλέψω το μέλλον όπω είπατε και εσεί. Αλλά αυτό που μπορώ να σα πω είναι ότι πρώτον έχουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο εκκινούμε τώρα για να δούμε πώ μπορούμε να επιτύχουμε, πώ μπορούμε να ασκήσουμε μεγαλύτερη επιρροή για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για ε, δοκιμές και θεραπεία. Πρόσφατα, πριν από μια εβδομάδα, είχα μια σχετική σύσκεψη πριν να έρθω εδώ και ο στόχος μας είναι να ολοκληρώσουμε κάτι το ουσιώδες μέχρι τα τέλη του 2020. Αυτά σχετικά με την πιθανή συμβολή μας. Δεν μιλούμε να μην μιλούμε δηλαδή μόνο για βέλτιστες πρακτικές, αλλά να, κάνουμε, να λάβουμε πραγματικές πρωτοβουλίες για να τις υποστηρίξουμε. Κάτι άλλο που εκκινούμε τώρα και που θα κορυφωθεί το χρόνο τον Οκτώβριο είναι κάνουμε προβλέψεις για το μέλλον προσπαθώντας να συντάξουμε μια μελέτη σε συνεργασία και με ορισμένα ε, Ινστιτούτα εταίρους για να, δρούμε, να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη τα επόμενα 10-15 χρόνια ορισμένων θεμάτων που έχουν άμεση σχέση με την κατάχρηση ναρκωτικών, ενδεχόμενη εξέλιξη νέων ψυχοτρόπων ουσιών, φεντανίνες και άλλα σχετικά με ναρκωτικά. Και το άλλο θέμα θα είναι πιθανότατα πώς μπορούμε να επηρεάσουμε μέσω και μακροπρόθεσμα την αντιμετώπιση δηλαδή των επιδημιών της υπαθήτητας ε, γάμα και να μην ξεχνούμε και τους οροθετικούς διότι αυτό που ε, με ανησυχεί ιδιαίτερα είναι ότι η γενεά αυτών που επινόησαν ήδη από τη δεκαετία του 80 τις ε, πρακτικές μείωσης του κινδύνου σιγά σιγά συνταξιοδοτούνται και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι επόμενες γενναίες ερευνητών θα συνεχίσουν την εργασία αυτή αποδίδοντάς της την ίδια σημασία ενώ βέβαια αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα και άλλες προκλήσεις. Αυτή η δουλειά ε, δηλαδή της παράδοσης της σκητάλης και της διασφάλισης ότι θα επιμείνουμε, θα εμείνουμε, θα βοηθήσουν να αντιληφθούν οι άνθρωποι ότι η γάμα Β και ε, το, ο ιός του AIDS δεν είναι κάτι που έχει ξεχαστεί στο παρελθόν διότι τότε υπήρχαν ε, τα προβλήματα αυτά ενώ σήμερα όχι. Υπάρχει το πρόβλημα και σήμερα αλλά είναι κάπως πιο κρυμμένο. Αυτά είναι δύο πράγματα για τα οποία όχι μόνο τα έχουμε περιλάβει στη στρατηγική μας για το 2025 αλλά υπάρχει και πραγματική δέσμευση ολόκληρου του οργανισμού μας του οποίου είμαι διευθυντής και το γεγονός ότι ως αποτέλεσμα της εφαρμογής στρατηγικής για πρώτη φορά τώρα το EMCDDA ως όργανο προστασίας δημόσιας υγείας εργάζεται για αυτές τις προτεραιότητες και για τις μολυσματικές νόσους βάζοντας αυτές τις προτεραιότητες. Και ε, το, η προθεσμία της, του ενδιάμεσου σταδίου είναι 2000, τέλος 2020. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ ενδιαφέρον. Ήμουν σίγουρη ότι οι συνάδελφοι θα έβρισκαν πολύ ενδιαφέρουσα την παρουσίασή σας και γι' αυτό σκέφτηκα να σας προσκαλέσω για πρώτη φορά όπως είπαμε ενδεχομένως να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με το κέντρο σας γιατί χρειάζομαστε δεδομένα και υπάρχουν ερωτήματα που τίθεται γνωρίζετε πολλά από αυτά τα θέματα. <clears throat> Όπως ήδη γνωρίζετε, τώρα θα περάσουμε στο θέμα της κάνοβης, για πάλι. Αν προκύψουν ερωτήσεις φυσικά για τη χρήση της κάνοβης ε, για ιατρικούς σκοπούς. Αυτό είναι το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης και σας ευχαριστώ πολύ. Uh, η συντάκτρια του αιτήματο, η κυρία Κονέτσουνα, δεν βρίσκεται εδώ. Υπάρχει αντικαταστάτης, η κυρία Τόρες. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να θέσω ένα θέμα πολύ σοβαρό ένα θέμα σοβαρό που σχετίζεται και με τα προηγούμενα. Μας ενδιαφέρει να δούμε πώς θα ε, σχολιάσουμε την νομοθεσία πριν εγκριθεί και θα ήθελα εδώ να αναφέρω το θέμα της χρήσης κάναβης γιατρικούς σκοπούς. Ε, να μην ξεχνάμε τον αφόρητο ανθρώπινο πόνο που προκαλούν ε, το AIDS, το Alzheimer, ο καρκίνος, χρόνιες παθήσεις ε, όπως η νόσος του Πάρκινσον ή η κατά Και από το 2017 ο ΠΟΗ θεωρεί ότι η κάναβη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς θεραπευτικούς για την επιληψία και τον αυτισμό. Αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ναρκωτικό, αλλά φάρμακο. Δηλαδή δεν ε, βλάπτει την υγεία, ίσα ίσα καταπολεμά την, ε, τον πόνο. Μετά από μήνες ε, ερευνών η κάναβης και το μόριο αυτό που αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία, της, ε, τα δύο βασικά στατικά της μαριχουάνας, μπορεί να αντιμετωπίσει τον πόνο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καλή υγεία ανθρώπων που αυτή τη στιγμή παίρνουν φάρμακα για να αισθανθούν καλύτερα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να νομοθετήσουμε τη χρήση της κάναβης μακροπρόθεσμα. Η θεραπευτική μαζική χρήση της κάναβης είναι γνωστή από καιρό. Οι δυτικέ κοινωνίες έχουν βέβαια στιγματίσει την ε, χρήση της κάναβης ακόμη και ιατρικούς σκοπούς και υπάρχουν ε, ασθενείς, ε, χρόνια ασθενείς, οι οποίοι ζουν το στίγμα αυτό ενώ απλώ θέλουν να κουφιστούν από τον πόνο του. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει και με θεμελιώδει ελευθερίε και με την ε, χρήση τη κάναβη και με μια σφαιρική προσέγγιση, την οποία θα πρέπει να την δούμε ε, σφαιρικά, ε, συνολικά. Δηλαδή και την αποπονικοποίηση ή ποινικοποίηση τη κάναβη και τι μέτρα θα ληφθούν. Στην Ισπανία πέρσι Ε, μας απασχόλησε το θέμα αυτό ε, και με καλλιέργεια κάναβης για θεραπευτικούς σκοπούς. Τα είπα, από 7 πολιτείες επιτράπει η χρήση της κάναβης και αυτό επέτρεψε να δημιουργηθούν και νέες θέσεις εργασίας. Ε, στην Ισπανία ε, η νομιμοποίηση μπορεί να καλύπτεται και από άδεια Γιατρικού σκοπού στην αγορά, δηλαδή κάναβη που παράγεται με τρόπο οικολογικό. Ή αν δούμε τις ε, απαιτήσει χωρών όπω το Ισραήλ τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει πρωταγωνιστέ στην έρευνα και ανάπτυξη και τη χρήση κάναβη για ιατρικού σκοπού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλά ήταν λοιπόν να αποδεχθεί την πραγματικότητα και να περάσει σε βήματα νομιμοποίηση τη κάναβη για ιατρικού σκοπού. Το Βέλγιο, η Αυστρία, η Δημοκρατία τη Τσεχία, η Μακεδονία, η Κροατία. Ε, και άλλες χώρες έχουν λάβει τα πρώτα απαραίτητα βήματα. Από τον Ιανουάριο φέτος και η Ελλάδα έχει κάνει μια παρόμοια κίνηση. Εάν λοιπόν εμεί δεν προλάβουμε την αγορά, η αγορά θα μας ε, προλάβει. Μεγάλες τράπεζες όπως η Κάισα και η Μπάνκτελ έχουν ε, ήδη μεγάλο κέρδος από τις πωλήσει κάναβης. Πρέπει να αυξήσουμε τις δυνατότητες της ιατρικής έρευνας και να προχωρήσουμε ε, συμφιλειωνόμενοι και με το ε, παρελθόν, με το τι απαιτήσει υπάρχουν από τους χρήστες, τους περιορισμούς που η φύση ίδια μας επιβάλλει, θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε τι δρόμοι ανοίγονται για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον και στην Νότια Ευρώπη και αλλού. Ευχαριστούμε πολύ και για την ανταλλαγή απόψεων εδώ. Θα μας μιλήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από την DG Home έχουμε την κυρία Ματζαρίνη, η οποία είναι διευθύντρια τη της πολιτικής για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο και τη διακίνηση ναρκωτικών. Έχετε το λόγο, κυρία Ματζαρίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την ανταλλαγή απόψεων ε, στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για, το χρήση, για την ε, χρήση της κάρβης για ιατρικούς σκοπούς. Πρέπει καταρχήν να ε, σας περιγράψω τους χώρους της δουλειάς μας τα κράτη-μέλη έχουν τη βασική αρμοδιότητα στα θέματα δημόσιας υγείας και σε σχέση με την βλάβη στην υγεία που έχει σχέση με τα ναρκωτικά. Εμείς ως Επιτροπή βοηθάμε, στηρίζουμε τα κράτη-μέλη στις αποφάσεις τους στο επίπεδο της πολιτικής τους σύμφωνα με το κοινοοικονομικό πλαίσιο. Η κάναβης υπό την έννοια αυτή αντιμετωπίζεται όπως, όλα τα υπόλοιπα, ε, ε, όπως όλες οι υπόλοιπες ουσίες. Έχουμε στην Γενική Διεύθυνση προσπάθειες μείωσης και πρόληψης και ένας άλλος τομέας στον οποίο εργαζόμαστε από την θέση ενισχύ της, του δεύτερου από τα δύο προγράμματα δράσης για τα ναρκωτικά που καλύπτει την περίοδο 2017-2020 που θα μας οδηγήσει στο τέλος της στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά. Παρακολουθούμε τι ε, συμβαίνει ε, στα μοντέλα ε, χρήσης της κάναβης και σε κράτη-μέλη και σε τρίτες χώρες, ώστε ενδεχομένως να αποκτήσουμε μια γενική εικόνα του τι ε, συμβαίνει. Ακριβώς ε, αυτό επεσήμανε και ο Διευθυντής του Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας. Υπάρχει παρακολούθηση, υπάρχει ε, ένα έντυπο το οποίο εκδόθηκε πέρυσι το 2017 από το Κέντρο Παρακολούθησης που αφορά την νομοθεσία της, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την Κάναβη. Θα υπάρχει και άλλη, και άλλο, και έκδοση. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε αυτή οι οποίοι θα λάβουν τι αποφάσει να, να ενημερωθούν. Αναφέρθηκα στην κάναβη ως ε, ναρκωτικό γιατί είμαστε στο πλαίσιο της στρατηγικής του πρόγραμμα δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για, ε, για τα ναρκωτικά. Όμως η ιατρική χρήση της κάναβη ξεφεύγει από αυτό το χώρο. Όσο περισσότερο χρησιμοποιείται η κάναβη για τι θεραπευτικέ της ε, ουσίε, γίνεται κανονικό φάρμακο και υπάρχει ένα λάθος νομοθεσίας να μιλάμε για φαρμακευτική κάναβη ή ε, ιατρικές, ε, κάναβη για ιατρικούς σκοπούς. Αλλά όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, εδώ μιλάμε για άλλο πράγμα, για τη φαρμακευτική χρήση ως φάρμακο δηλαδή, που είναι αυτό το οποίο παρακολουθούμε. Η συζήτηση έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, εξακολουθεί το θέμα να είναι αμφιλεγόμενο, Επίση αντιλαμβάνομαι και από αυτά που δημοσιεύονται στον τύπο, η κάναβης ε, για ιατρικούς σκοπούς όπως ήδη περιγράφεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Αυστραλία και σε κάποια κράτη-μέλη περιλαμβανομένου και του δικού μου της Ιταλίας, η κάναβης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θεραπευτικούς λόγους, κυρίως όταν αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει άλλη ε, θεραπεία που μπορεί να ανακουφίσει χρόνιους πόνους ε, ή άλλες καταστάσεις όπως η επιληψία, ο καρκίνος και άλλα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να εργάζεται στο χώρο της συγκέντρωσης των απαραίτητων πληροφοριών. Θα μας πείτε ενδεχομένως ότι υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες, αλλά εξ όσων γνωρίζουμε υπάρχουν εξαιρετικά αξιόλογες αναφορές που λένε ότι πρέπει να προχωρήσουμε, ε, έπρεπε να είχαμε, το είχαμε ήδη κάνει, ε, να είχαμε προχωρήσει ε, για την έγκριση για ιατρικούς σκοπούς και εξίσου σημαντικές εκθέσεις που μας λένε ότι η τεκμηρίωση που έχουμε δεν είναι επαρκής. Βρισκόμαστε προς το παρόν σε ένα δίλημα και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο αναλύουμε και παρακολουθούμε την κατάσταση όπως κάναμε τα τελευταία χρόνια και όπως θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα οι συνάδελφοι που θα ήθελα να πάρουν τον λόγο. Επ' αυτό, η κυρία Ιούσο. Eh, Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. δεν θα επιχειρηματολογήσω κατά των όσων ακούσαμε, διότι δεν μπορώ πραγματικά για το κατά πόσο είναι ναρκωτική ουσία η φαρμακευτική κάναβη. Όμως έχω ένα γνωστό, ευρωβουλευτή μάλιστα, ο οποίος υποφέρει από μια χρόνια πάθηση. Υποφέρει μάλιστα πάρα πολύ και έχουμε συζητήσει για, τη χρή... για την ανάγκη να χρησιμοποιεί κάναβη οι ιδιότητες της κάναβης. Και έχει μια ε, σειρά από τέτοιες ευνοϊκές ιδιότητες, θεραπευτικές ιδιότητες, ε, είναι γνωστές, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι υπάρχει και αντίλογος. Όσες καλές ε, επιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν, μπορεί να υπάρχουν και οι αντίθετες. Πάντως, για τη χρόνια πάθηση πρέπει να δούμε τι Συνέπειε μπορεί να υπάρχουν από αυτό και σκοπιά, γιατί σε πολλού δίνουν ηρεμιστικά, παυσίπονα, πολύ ισχυρά. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει η κατάλληλη έρευνα και την ανάλογη ε, ενδελεχή έρευνα να κάνουμε και για την ίδια την κάναβη και το τι χρήση μπορεί να έχει. Χρειάζονται πόροι επίσης. Χρειάζεται να διατεθούν πόροι γιατί ακούσαμε ότι υπάρχουν πολλές μελέτες, πολλές είναι υπέρ της χρήσης της κάναβης για ιατρικούς σκοπούς αλλά το θέμα είναι κατά πόσον πρόκειται για σοβαρέ μελέτε ή απλώ μια αξιολόγηση. Κάποιοι που λέει ναι, πήρα λεγικά κάναβη και στάθηκα καλύτερα. Αλλά μπορεί να υπάρχουν, δευτερο... να υπάρχουν παρενέργειε τι οποίε δεν γνωρίζουμε. Είναι λοιπόν σημαντικό να γίνει έρευνα ενδελεχή, επιστημονική, να δούμε όλε τι ε, εξονυχιστικέ λεπτομέρειε του θέματο και το κατά πόσον μπορεί η κάναβη να χρησιμοποιηθεί πραγματικά για ιατρικού σκοπού, σε τι ποσότητε και πώ μπορεί να χρειάζεται να απομακρυνθούμε από τις σημερινές πρακτικές της ε, αυτοθεραπείας κάποιων ανθρώπων ε, που χωρίς την παρακολούθηση που χρειάζεται από γιατρό παίρνουν ό,τι να Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ντάλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ επίσης και την κυρία Ματσαρίνη για τη συζήτηση του πολύ σημαντικού θέματος. Αυτό που συζητάμε σήμερα εδώ είναι η κάναβης ε, που χρησιμοποιείται για ιατρικούς σκοπούς. Το υπογραμμίζω αυτό γιατί η αφετηρία είναι ότι δεν μπορούμε να συγχαίουμε τη συζήτηση ε, για τις κάναβες για ιατρικούς σκοπούς με την ψυχαγωγική της χρήση. Αυτό είναι μια σύγχυση που γίνεται πάρα πολύ συχνά. Ακόμα και αν δούμε το νομικό σκέλος και τον κανονισμό, βλέπουμε ότι πρόκειται για δύο τελείως διαφορετικά θέματα, εντελώς χωριστά μεταξύ τους. Ε, η συζήτηση για ιατρικούς σκοπούς πρέπει να επικεντρώνεται αποκλειστικά για προϊόντα που κατασκευάζονται σε ελεγχόμενο και ε, ρυθμιζόμενο περιβάλλον. Ε, ε, υπάρχει θέμα ειχνηλασιμότητας και ασφάλειας και όταν εξασφαλιστούν αυτά το επόμενο βήμα είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ίση πρόσβαση των ασθενών σε αυτή. Γιατί τελικά τι νόημα έχει η ρύθμιση αν μόνο λίγοι έχουν πρόσβαση σε αυτού του είδου το φάρμακο. Η έρευνα όπως ήδη ακούσαμε είναι στο επίκεντρο όλων. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνουν διαφορετικές μελέτες ε, επί διαφορετικών θεμάτων της ε, ΚΑΜ. Έχει πάνω από 130, υπάρχουν 130 διαφορετικά καναβιοειδή ε, που είναι το 40% των φυτών. Αναφερθήκαμε στο λάδι CBD που είναι πολύ αποτελεσματικό σε περιπτώσεις πόνων όπως η Πάρκινσον και η σκλήρινση κατά πλάκας και πολλές άλλες παθήσεις. Και συνεχίζεται η έρευνα για την ιατρική χρήση της κάναβης σε άλλες παθήσεις, άρα πρέπει να συγκεντρώσουμε περισσότερες πληροφορίες και να μάθουμε πολύ περισσότερα. Είναι ευπρόσδεκτες λοιπόν οι προσπάθειες που γίνονται σε διάφορα κράτη-μέλη. Ανακούσαμε ε, πολλά ε, ε, κράτη-μέλη. Ακούσαμε ότι στι ΗΠΑ και του Ισραήλ γίνονται προσπάθειες και οι εξελίξεις και στη Μάλτα, τη χώρα μου, για την διερεύνηση του σενάριου προς αυτήν την κατεύθυνση. Ελπίζω ότι οι εξελίξεις αυτές θα βοηθήσουν την ε, ενίσχυση της έρευνας στον τομέα αυτό Πιστεύω ότι το δίκτυο ανταλλαγή ευρημάτων, νέων, νέων ευρημάτων και βέλτιστων πρακτικών μπορεί να αναπτυχθεί ανάμεσα στου ερευνητέ για να δουν τι είναι αποτελεσματικό, τι μπορεί να γίνει. Και θέλω ε, να κάνω κάποιε ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέμα τη εξασφάλιση καλύτερη ποιότητα και περισσότερη έρευνα από αυτού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πρόθυμη να χρηματοδοτήσει ε, την ε, περαιτέρω έρευνα ώστε να την Και επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πρόθυμη να ζητήσει ε, ε, ε, στην Ευρωπαϊκή Αρχή Φαρμάκων για κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τον την ελεγχόμενη χρήση κάναβης και σκοπεύει να δουλέψει, να εργαστεί για έναν κανονισμό και την ίση ε, πρόσβαση στα φάρμακα που στηρίζονται ε, στην κάναβη σε όλη την Ευρωπαϊκή ε, Ένωση και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ναρκωτικών και Τοξικομανίας που δημοσιεύουν εκθέσεις κάθε λίγους μήνες, θα ήθελα να ξέρω αν, λαμβάνετε, αν πραγματικά πραγματοποιείται έρευνα στον τομέα. Ευχαριστώ κύριος Φλάναγκαν. Ως είπε και η προλαλήσασα, είναι σημαντικό να διαφοροποιήσουμε ανάμεσα στην χρήση της κάναβης για ψυχαγωγικούς και για ιατρικούς σκοπούς. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάπως δεν πήγε πολύ καλά εδώ κατά τη συζήτηση του θέματος, γιατί πολλά από αυτά που αναφέρατε δεν έχει σχέση με την ιατρική χρήση, ήταν οτιδήποτε άλλο. Εμείς επειδή αναφέρθηκαν πολλές χώρες, η Ιρλανδία φέτος έχει δώσει άδεια σε κάποιους να χρησιμοποιήσουν την κάναβη για ιατρικούς σκοπούς. Αλλά αυτό, γι' αυτό χρειάστηκαν τεράστιες μάχες από αυτούς οι οποίοι χρειάζονταν την πρόσβαση σε αυτό το φάρμακο. Μία συγκεκριμένη κυρία, η οποία το μιλάει δημόσια, είναι και φίλη μου, η Βίρα Τούμι, και αυτό σχετίζεται με αυτό που είπαμε για το CBT και την ιατρική για, τα, ε, για τις ουσίες που προέρχονται από την κάναβη, ε, πάσχει από το σύνδρομο Τραβέτ ε, από τη στιγμή ε, ξόδευε 150.000 ευρώ το χρόνο σε νοσηλεία, να μην από τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η κόρη της μπορεί κανείς ε, και στην Ιρλανδία και σε πολλές άλλες χώρες ε, να έχει ε, πρόσβαση στο CBD που δεν είναι η ψυχοδραστική ουσία. Αλλά όταν μιλάμε για το σύνδρομο ΤΕΒΕΤ η ουσία που χρειαζόταν ήταν άλλη και δεν υπάρχει πρόσβαση σε αυτή χωρίς άδεια. Η κυρία αυτή τώρα πρέπει να πάει στην Ολλανδία κάθε τρει μήνες και να πληρώσει ένα σωρό λεφτά για να επιστρέψει με το φάρμακό της. Πρέπει να, αλλάξει αυτή η κατάσταση γιατί από τη στιγμή που ω παιδεία να παίρνει το φάρμακο πλέον δεν, υπάρχει, δεν έχει καμία κρίση. Καμία κρίση. Πρέπει να γίνουν μελέτες. Είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει μελέτη αν δεν ήταν έγκλημα η κατοχή. Αλλά γνωρίζουμε σε, από πάρα πολλές περιπτώσεις ότι άλλαξαν ζωές ανθρώπων. Πρέπει λοιπόν να κινηθούμε από αυτού και ο μόνος τρόπος να προχωρήσει το θέμα είναι σαφώς να γίνει διάκριση ανάμεσα στην ιατρική και τη μη ιατρική χρήση. Κάτι πρέπει να κάνουμε από αυτού γιατί τώρα αντιμετωπίζουμε πρόβλημα αυτή την κυρία στην Ιρλανδία. Μας λένε ότι θα ήταν παράνομο το κράτος να ε, το εισάγει επισήμως από την Ολλανδία. Προτείνεται στην ε, οικογένεια να μεταβεί στην Τσεχία γιατί εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα νόμιμης εισαγωγής. Και τώρα τίθεται το θέμα. Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ποια είναι η συνεκτικότητα, η συνέπεια που υπάρχει στα προϊόντα. Το παιδί αυτό έχει τρομοκρατηθεί και φοβάται ότι παρότι η ουσία πάει πάρα πολύ καλά ε, αυτή από την Ολλανδία φοβάται ότι η αλλαγή σε ένα πάλο προϊόν που παράγεται από μια άλλη εταιρεία μπορεί να μην είναι εξίσου καλή, καλά το αποτέλεσμα. Με, ε, έρχονται σε επαφή μαζί μου εκατοντάδες άνθρωποι που πραγματικά περνάνε από, το, από, το, δυσκολίες. Υπάρχει κάποιος ο οποίος πρέπει να φοράει ε, ε, πάνες ακράτειας αν δεν χρησιμοποιεί αυτού την κάναβη. Οι άνθρωποι περνάνε από πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες και το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά αν βοηθάνε τους, βοηθάει τους ανθρώπους πρέπει η πρόσβαση των ανθρώπων, ε, ναι, ε, πρέπει ε, να, να, υπάρχει πρόσβαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το μικρόφωνο πάλι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω είχατε εξής μια ερώτηση για τον Διευθυντή κ. Γκουστίλη. Πρώτα εσάς. Εσείς και Γκουστίλ παρακαλώ να απαντήσετε. Μετά η κυρία Μοζερίνη της Επιτροπής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους και όλους ημών για τα σχόλια και τις παρεμβάσεις σας. Τα περισσότερα από τα σχόλιά σας είναι πάρα πολύ σημαντικά και αποτελούν σημαντική συμβολή στο έργο μας. Πρώτα, το EMCDDA για την ώρα έχει αναθέσει την επανεξέταση των εκθέσεων για τη θεραπευτική αξία της κάναβης, σχετικά δηλαδή με την αξιολόγηση των ενδείξεων, και θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να ε, δημοσιεύσουμε τη σχετική έκθεση πριν από τα Χριστούγεννα φέτος, με την ιδέα να συλλέξουμε όσο το δυνατόν περισσότερες μελέτες και εκθέσεις είναι δυνατόν και να έχουμε και την υποστήριξη διεθνών εμπειρογνωμόνων για να μας εξηγήσουν τι μπορούμε να πούμε και ποιες θα πρέπει να είναι οι ιδιότητες που θα πρέπει να προσέχουμε του προϊόντος αυτού. Τονίζω ότι προέτους η Αμερικανική Ακαδημία Τεχνολογίας κλπ. μίλησε για, την, για τις θεραπευτικές ιδιότητες της κάναβης, ε, κάτι το οποίο ελέγχθη και είναι και ένα από τα θέματα που θα ήθελα να τονίσω και εγώ, είναι ότι Εάν εξετάσει κανείς τη γνώση που έχουμε σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για τις θεραπευτικές ιδιότητες της κάναβης, θα δούμε ότι βρισκόμαστε λίγο πολύ στην ίδια θέση σχετικά με τα όσα γνωρίζαμε και με τα neurotransmitters πριν από 20 χρόνια. Να γνωρίζουμε ότι εάν δεν επενδύσει κανείς στην έρευνα δεν πρόκειται να κατανοήσει ποτέ καλύτερα ποιες είναι οι ιδιότητες και οι δυνατότητες των ε, προϊόντων της κάναβης. Νομίζω η κυρία Ντάλη είπε ότι και μια από τις ουσίες που περιέχει μάλλον η ίδια η κάναβη είναι σημαντική και γι' αυτό στο MCDDA δεν μας αρέσει τόσο πολύ να χρησιμοποιούμε τον όρο ιατρική κάναβη διότι δεν μιλούμε και για ιατρικό όπιο, μιλούμε για θεραπεία ασθενών με μορφήνη, για παράδειγμα σε περιπτώσεις καρκινοπαθών. Επανέρχομαι στα σχόλια του κ. Φλάναγκαν. Επειδή δεν γνωρίζουμε τις πραγματικές ιδιότητες κάποιων από τα εκχυλίσματα αυτά και δεν έχει γίνει αρκετή έρευνα για αυτά, θεωρώ ότι ενδέχεται να βρισκούμε να βρεθούμε στην ίδια θέση όπως και προ 25 ετία. και σε ορισμένε χώρες δεν έχουν προχωρήσει τα πράγματα. Υπάρχουν μάλιστα περισσότερα εμπόδια και ε, για τη χρήση της κάναβης για καρκινοπαθή παιδιά. Γιατί φοβούνται πολύ ότι μπορεί τα παιδιά να γίνουν τελικώς ε, τοξικομανείς. Χρειαζόμαστε λοιπόν σαφώς πολύ περισσότερες ενδείξεις για να καταλήξω με κάποιο πιο θετικό και επικοδομητικό τόνο, Κάτι που είναι ενδιαφέρον είναι εάν το παρόν Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να προσθέσουν μια προτεραιότητα για τα μελλοντικά ερευνητικά προγράμματα μεταξύ αυτών και όσα θα συζητήσετε στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για τον προπολογισμό της Ένωσης, να περιλάβετε και αυτά τα πράγματα, διότι είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει επαρκής έρευνα και χρειαζόμαστε ένα μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα και για αυτά. Το ίδιο όπως έχει γίνει για παράδειγμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν θα δούμε την κάναβη σαν κάτι καλύτερο από τη μορφήνη, διότι πράγματι υπάρχουν καταστάσεις ανθρώπων όπου η χρόνια χρήση των οπιοειδών έχει τελικά δυσμενείς επιπτώσεις στη υγεία τους και ίσως μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις η κάναβική να βοηθούσε έστω και αν δεν έχει την ίδια ε, επίδραση όπως ε, για παράδειγμα η μορφίνη. Και τέλος δεν είναι μονάχα η κάναβης, υπάρχουν και άλλες ουσίες που μπορούν να έχουν θεραπευτικό αποτέλεσμα. Διεξάγεται στις ΗΠΑ μελέτη για την χρήση του MDMA που είναι το όνομα του έκσταση για την αντιμετώπιση μετατραυματικών ε, διαταράξεων. Νομίζω ότι αν γίνει μια σχετική έρευνα, ίσως σε 10-15 χρόνια να μην ακούμε πλέον μαρτυρίες σαν αυτές που ακούσαμε σήμερα. Ευχαριστώ κυρία Μοτσαρίνη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να απαντήσω στις ερωτήσεις της κυρίας Ντάλη. Νομίζω κανείς δεν αρνείται ότι είναι θεμελιώδης η έρευνα και μελέτη ως προς τα θέματα αυτά και χρειάζεται να υπάρξει και απαραίτητη επένδυση πόρων για να γίνει σωστή έρευνα. Δεν είμαι σε θέση να σας δώσω συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς θα χρησιμοποιηθούν κονδύλια για αυτό το σκοπό. Πάντω, εφόσον προβλεφθεί στην ημερήσια διάταξη άλλη επιτροπή, ευχαρίστω να σα δώσουμε περισσότερε λεπτομέρειε για τα στοιχεία τη χρηματοδότηση όλου αυτού του θέματο. Το ίδιο και για τι κατευθυντήριε γραμμέ. Εάν ληφθεί κάποια απόφαση από κοινού, από το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα και ότι μπορούμε να δουλέψουμε μαζί όλοι για να προχωρήσει το θέμα αυτό, θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερη πρόοδο στη δουλειά μας. Πάντως υπάρχουν πολλές μελέτες που λένε κάτι και μετά υπάρχουν αυτές που λένε και το αντίθετο. Υπάρχουν στοιχεία των ΠΟΗ με έρευνες που γίνονται από χρόνια για την κάναβε ιατρικούς σκοπούς. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απλώς δεν μπορεί παρά να λάβει υπόψη όλο τον πόνο και την οδύνη που υπάρχει γύρω μας και που ενδεχομένως να μπορούσε να ε, θεραπευθεί, να ανακουφιστεί με τη χρήση κάναβης γιατρικού σκοπούς, αν αποδειχθεί η πραγματική αποτελεσματικότητα των προϊόντων αυτών με πραγματική έρευνα ε, και βεβαιωθούμε ότι υπάρχουν μόνο ωφέλη και όχι παρενέργειες και ένα μετριασμένο κόστος, θα προχωρήσουμε. Αυτά είχα να πω προ στιγμή. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ όλου του συναδέλφου για τη συμμετοχή του στην ε, συζήτηση αυτή. Ε, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα ε, που πρέπει να το προβλέψουμε στην ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την κυρία Μοτσαρίνη και τον κύριο Γκροστέλ που συμμετείχε. Και τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Αντίρρηση, αντιρρήσεις μάλλον. Δύο αντιρρήσεις. Για γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. Νομίζω τα έχετε στους φακέλους σας, δεν θα το διαβάσω τώρα, δεν χρειάζεται να διαβάσω τους αριθμούς. Καλαμπόκι είναι. Οι αντιρρήσεις αρκετών από τους συνεισηγητές είναι δύο ε, βασικά που θα μας αποσχολήσουν σήμερα, γιατί υπάρχουν και άλλες. Και μετά το λόγο θα έχουν οι συνάδελφοι που θέλουν να παρέμβουν. Ε, εκ μέρους του κυρίου Στάς, η κυρία Χέμπιχ. Ευχαριστώ, λέγομαι Χόιμπουχ. Είμαι συνάδελφος του Μπατστάς και συνεργάζομαι μαζί του σε άλλε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ. Ο Δε Μπάρτ με παρακάλεσε σήμερα να τον αντικαταστήσω, διότι είναι απασχολημένο, είναι στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού, όπου καταθέτει 35 εκθέσει απαλλαγή. Και γι' αυτό το λόγο ε, αντιλαμβάνεστε ότι κολλείεται. Μιλούμε σήμερα για δύο αντιρρήσει, ενστάσει κατά της ε, κυκλοφορίας δύο γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Τις ε, ενστάσεις αυτές καταθέτουν ο Μπάρτ και άλλοι πέντε ευρωβουλευτές. Πρόκειται για τροποποιημένο ε, καλαμπόκι, το ΜΟΝ 47 και άλλα δύο τροποποιημένα προϊόντα και για το καλαμπόκι 59-12 όπου η Επιτροπή Περιβάλλοντος έχει λάβει 22 ενστάσεις. Τέσσερις από αυτές αναφορικά με την καλλιέργεια των προϊόντων αυτών στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες 18 για τις εισαγωγές ε, τροφίμων. Πέραν των δύο αντιρρήσεων ενστάσεων που συζητούμε σήμερα, όλες οι υπόλοιπες έγιναν δεκτές στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να επιτρέπει συστηματικά την εισαγωγή ε, γενετικώς τροποποιημένων προϊόντων χωρίς να λαμβάνει υπόψη την γνωμοτήση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί προσβολή κατά των Ευρωπαίων ε, πολιτών. Οι ενστάσεις ε, μάλλον υποτίθεται ότι αυτά έχουν ανθεκτικότητα σε γλυφοσάτη και γλυφοσινάτη. Αυτά όμως θέτουν ερωτήσεις για την ασφάλεια των καταναλωτών. Δεν υπάρχει επαρκής αξιολόγηση του κινδύνου που θεμελιώνεται και με πολλές κριτικές παρατηρήσεις των αρμοδιών αρχών των χωρών μελών σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση κινδύνου της ΕΦΣΑ. Δεν λαμβάνεται υπόψη η αρχή της προφύλαξης, καθώς και μεμφόμεθα, μάλλον για μη δημοκρατική διαδικασία λήψη αποφάσεων. Για τα άλλα προϊόντα, 87, 427 και μόνο 89, 89-34 και επίσης το 87, 427 που ε, διασταυρώνεται με το 89, 034 και το NK603, δεν έχουν υποβληθεί σχετικές αιτήσει από την Μονσάντο. Ενώ η ΕΦΣΑ θεωρεί ότι τα προϊόντα αυτά είναι ασφαλή, χωρίς να γίνει αξιολόγηση κινδύνου όλων των υποσυνδυασμών, δεν μπορεί να θεωρηθεί πλήρης. Για το καλαμπόκι αυτό έχει γίνει ανθεκτικό κατά της γλυφοσυνάτης λόγω της τοξικότητάς του από τον Ιούλιο του 2018 δεν επιτρέπεται πλέον η χρήση του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέθεται όμως τότε το ερώτημα πώς είναι δυνατόν ένα ριζανιοκτόνο που είναι υπερβολικά τοξικό για να χρησιμοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να εισάγεται μέσω του ε, γενικά τροποποιημένου καλαμποκιού η ΕΦΣΑ δεν αξιολογεί τα κατάλοιπα των ζυζανιοκτώνων. Ούτε υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το εάν κατάλοιπα γενετικά τροποποιημένων ανθεκτικών ζυζανιοκτώνα φυτών εμπίπτουν στις ε, διατάξεις περί ανώτατων ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την έκθεση του 2015 της ΕΦΣΑ για κατάλοιπα ζυζανιοκτώνων, δεν αποδίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις, στα φυτά χρήσης εισαγόμενα. Παρόλο που από τη φύση τους έχουν περισσότερα κατάλοιπα ζυζανιοκτώνων από μη τροποποιημένα φυτά. Το ψήφισμά μας απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην επιτρέπει εισαγωγές γενετικά τροποποιημένων ε, φυτών για τα οποία στην Ευρωπαϊκή Ένωση μάλλον τα οποία είναι ανθεκτικά σε ζανιοκτώνα τα οποία είναι απαγορευμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω έλλειψης επαρκών ενδείξεων και πληροφοριών σε αυτή τη μία περίπτωση. Λόγω της ελλείψεως δεδομένων και των κενών στις γνώσεις της περιπτώσεις αυτές, το απαγορεύει η ε, απλή λογική. για να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας των κατανοητών. Στο όνομα του Μπατ ευχαριστώ τους συναδέλφους για την υποστήριξή τους της ενστάσεις κατά γενετικά τροποποιημένων οργανισμών που έχουμε υποβάλει στο παρελθόν και ελπίζω ότι την ίδια στάση θα τηρήσετε και αύριο στην διάρκεια της ψηφοφόρειας. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Εύη. κυρία Καντέμπαρ. Είστε έτοιμοι και μετά κυρία Εύη. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε που καθυστέρησα λίγο. Μιλάμε για το ε, Ναραβός το 87, 427 και το ε, 87, ε, 59-122. Το ένα αφορά ε, ε, την ε, αντοχή στο γλυφοσάτ και το άλλο στο γλυφοσυνικό αμμόνιο. Ε, οι δύο τροποποιημένοι γενετικά οργανισμοί αραβοσίτου είναι ε, ανθεκτικοί στο γλυφοσάτι ή το γλυφοσινικό αμμόνιο. Ο σκοπός είναι της αντιμετώπισης του προβλήματος των ε, ζυζανίων που αντέχουν στα φυτοφάρμακα σε διάφορες χώρες. Όμως ε, τα επολύματα των ψεκασμών δεν έχουν αξιολογηθεί και τα, υπεροχή, ε, και τα ε, επιχειρήματα στο παρελθόν έχουν, ε, έχουν ε, αναφερθεί σε παραμονή τους στις τροφές. Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση κινδύνου της ΕΦΣΑ για το mon 427 είναι ότι δεν θα πρέπει να είναι αποδεκτό επειδή δεν υπάρχουν δεδομένα για την πιθανή τοξικότητα και τις επιπτώσεις στο ανοσοποιητικό σύστημα. Επιπλέον, μια μελέτη δείχνει ότι οι υποθέσεις που αφορούν την μελέτη μελών, την ε, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι ανεπαρκής και ε, το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν τα απαραίτητα δεδομένα. Όσον αφορά τι προηγούμενε και αντιρρήσεις, θεωρούμε ότι δεν είναι σωστό η Κομισιόν, ενώ αναγνωρίζει την ύπαρξη σοβαρών προβλημάτων για την δημοκρατική νομιμοποίηση τη δικαστήρια λήψη αποφάσεων που αναφέρεται και στην επεξηγηματική έκθεση, στην αιτιολογική έκθεση, συνεχίζει να ε, προτείνει την έγκριση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών οργανισμών. Όλες οι προτάσεις ε, για την έγκριση αυτών των οργανισμών από την Κομισιόν δεν έχουν δώσει γνωμοδότηση ε, της Επιτροπής και έχουν οδηγήσει σε κατηγορική απόρριψη από το Κοινοβούλιο. Ο, ο κανονισμός 182 του 2011 αναφέρει ότι όταν λαμβάνουμε υπόψη μα τι επιπτώσει άλλων ε, ουσίων, κυρίως σε τομεί, την ε, φορολογία, την ασφάλεια των καταναλωτών και την προστασία του περιβάλλοντο, η ισόρροπη λύση θα πρέπει να προέρχεται με την αποφυγή οποιασδήποτε επικρατούσας άποψης που θα αφορά κάποια εκτελεστική πράξη. Παρά τα αυτά, η Κομισιόν συνεχίζει να εγκρίνει διάφορες ε, ποικιλίε γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, πράγμα που είναι ανάρμοστο και αντίθετο με την αρχή της ε, ε, πρόληψης. Κυρίως όταν είναι προφανές ότι οι προτάσεις δεν στηρίζονται ποτέ από τις απόψεις των κρατών μελών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τώρα η κυρία Εύη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να υποστηρίξω αυτήν την αντίρρηση που συνυπέργαψα με τους συναδέλφους. Μιλάμε για μια πολλωστή περίπτωση όπου στην αρμόδια επιτροπή για την τροφική λυσίδα των ε, έμβιων ζώντων και της ε, καλής τους υγείας δεν ε, έφτασε μια πιστική γνωμοδότηση. Και στις δύο υποθέσεις που μας απασχολούν σήμερα, τα γενετικώς τροποποιημένα καλαμπόκια. Τα κράτη-μέλη που ψήφισαν υπέρ της χρήσης τους στις σχετικές επιτροπές δεν είναι πλειοψηφία του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Αυτά τα δύο γενετικώ τροποποιημένα λοιπόν και δεν θα επεκταθώ γιατί οι συνάδελφοι εξήγησαν επαρκώς γιατί προβάλλουμε αυτή την αντίρρηση για την εξουσιοδότηση αυτών των νέων γαματαφόμικρων ή τέλος πάντων την επανεξουσιοδότηση των υπαρχόντων γαματαφόμικρων. Η πρώτη υπόθεση, το πρώτο καλαμπόκι της Μονσάντο το 87427 και Ε, το 89-034 είναι ε, ανθεκτικά στην γλυφοσάτη. Και όπως ήδη έχει διαπιστωθεί και έχει εξακριβωθεί από τα ε, στοιχεία, είναι ένα ζυζανιοκτόνο που χρησιμοποιείται σε δόσεις ένα και μεγαλύτερες και πιο ευρέως. Μπορεί να είναι και καρκινογενές. Πρέπει να δούμε λοιπόν τα κατάλοιπα του φυτοφαρμάκου αυτού στις οδιές γιατί είναι ένα θέμα που οπωσδήποτε πρέπει να εξεταστεί σοβαρά. Η αξιολόγηση αυτού του πρακτικού προβλήματος δεν έχει γίνει καθόλου όπως θα έπρεπε, για να μην πω ότι τελείως αγνοήθηκε. Δεν μπορούμε να το παραγνωρίζουμε λοιπόν. Επιπλέον δεν ελήφθη υπόψη η περαιτέρω δυνατότητα συνδυασμού αυτών των αραβοσίτων, διότι η εταιρεία Μονσάντο, Μονσάντο δεν έδωσε τα απαραίτητα δεδομένα, τα στοιχεία των πειραμάτων. Οπότε η ΕΦΣΑ θεώρησε ότι δεν υπάρχει κίνδυνο. Ε, κατά τη δική μου την άποψη, δεν μπορούμε έτσι να προστατεύσουμε την ε, υγεία των Ευρωπαίων πολιτών. Στη δεύτερη υπόθεση έχουμε την περίπτωση του Καλαμποκιού που έχει ένα θεκτικό στο, στην Γλυφοσυνάτη, Το Καλαμπόκι 59-122. Η εξοδότηση του θα εκπνεύσει μέσα σε ένα εξάμεινο. Μου φαίνεται λοιπόν ότι δεν μπορούμε να επανεγκρίνουμε κάτι που θα πάψει να χρησιμοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν δημοκρατικέ διαδικασίε και σχετικέ αποφάσει με τα γάματα όμικρον πρέπει να καλύψουν τις ανάγκες μας. Με την αναθεώρηση του κανονισμού θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην εγκρίνει αυτά τα καλαμπόκια, ε, να μην επιτρέψει να κινδυνεύσουμε σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν έχει την απαραίτητη γνωμοδότηση. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα οι σκιώδεις Ο κύριος Φιέλνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν πρέπει να αρχίσουμε με το ερώτημα τι ακριβώς κάνουμε εδώ και για ποιο λόγο έχουμε αυτές τις αντιρρήσεις. Οι αντιρρήσεις ενδεχομένως δεν είναι πολύ σημαντικό εργαλείο από νομική άποψη, γιατί δεν θα αλλάξουν και πάρα πολλά στην πράξη, αλλά έχουν σημαντική θεσμική λειτουργία. Είναι το εργαλείο που έχει το Κοινοβούλιο για να ελέγξει την Κομισιόν και αφορά τη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Και πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και να τα αντιμετωπίζουμε και πολύ προσεκτικά. Όταν έχουμε τέτοιου είδους περιπτώσεις ενώπιόν μας, αν πρέπει να δώσουμε μία αντίρρηση, θα πρέπει να εκπληρώνει τουλάχιστον ένα από τα εξής δύο κριτήρια. Πρώτον, θεωρούμε ότι η Κομισιόν έχει ξεπεράσει την εντολή της, δεν, έχει, δεν συμμορφώνεται με την ομοθεσία, δεν υλοποιεί την απόφαση σωστά. Και δεύτερο κριτήριο είναι αν πραγματικά είχαν παραβλέψει, αγνοήσει την επιστήμη. Τα επιστημονικά δεδομένα κάνουν κάτι παρότι η επιστήμη λέει το ακριβώς αντίθετο. Όσον αφορά το πρώτο κριτήριο, ότι η Κομισιόν δηλαδή αν ε, λειτουργήσε εντός ή εκτός του νόμου, δεν άκουσα κανέναν ούτε καν να ε, αναφέρεται ακροθυγός ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει. Ο τρόπος ε, συμμορφώνονται με αυτά που είπαμε. Μπορεί να μην μας αρέσει αυτό που κάναμε, αλλά αυτό έκαναν. Και το άλλο κριτήριο είναι αν ακολούθησαν τις συμβουλές της επιστήμης. Γιατί είναι θέμα επιστήμης. Εδώ γνωρίζετε ότι δεν είμαι ειδικό σε γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, ένα πράγμα γνωρίζω. Κανένας άλλος συνάδελφος δεν είναι παρκός ειδικό τουλάχιστον για να κρίνει αν και κατά πόσον είναι ασφαλές ή όχι επιστημονικά. Η νομοθεσία όμως αυτό το ε, έργο το έδωσε στην ΕΦΣΑ. Εμείς είπαμε στην ΕΦΣΑ, μήπως μπορείτε να δημιουργήσετε τα καλύτερα σώματα επιστημόνων που έχουμε. Το έκαναν, το έλεγξαν και είπαν ότι οι δύο αυτοί οργανισμοί γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί είναι όσο ασφαλείς, όσο και η συμβατική ομόλογή τους, έτσι είπαν. Αυτή τη στιγμή αρχίζω να μπερδεύομαι. Γιατί αντιστρέφονται τα πράγματα. Τώρα η συζήτηση εδώ αφορά. Ωραία μου θυμίζει ε, τη συζήτηση για την κλιματική αλλαγή που είχαμε για ένα διάστημα. Κάποια ε, συναδελφοί, ας πούμε, από το UKIP είπαν «Α, δεν έχουμε το είδος της κλιματικής αλλαγής που ισχυρίζεται ότι έχουμε για διάφορους λόγους και ότι τα επιστημονικά δεδομένα που μας υποβάλλονται είναι ελαττωματικά και υπάρχουν και άλλοι επιστήμονες, στους οποίους εγώ ήρθα σε επαφή και λένε άλλα πράγματα. Τώρα όμως ε, έχουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα ε, και αυτό συμβαίνει μερικές φορές γιατί γίνεται, ε, το, το εγκρίνει η πλειοψηφία της Επιτροπής. Το θέμα είναι ότι έχουμε την πιο αυστηρή νομοθεσία στον κόσμο για γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, τον πιο αυστηρό έλεγχο στον κόσμο και αυτοί οι δύο οργανισμοί πέρασαν από ακριβώς το μάτι της βελόνας. Πέρασαν αυτόν τον έλεγχο, αλλά παρόλα αυτά δεν τους θέλουμε ή τουλάχιστον η τάση είναι η πλειοψηφία της Επιτροπής να μην τους θέλει. Νομίζω ότι είναι κατάχρηση του, ε, η ε, κακη χρηση του νομικου αυτου μεσου σαφως υπονόμευσης της αξιοπιστίας των θεσμικών οργάνων που εμείς δημιουργούμε για να εργαστούν για μας και υπονομεύεται μια πολιτική που στηρίζεται σε επιστημονικά στοιχεία. Ελπίζω ότι περισσότεροι συνάδελφοι θα αμφισβητήσουν τον τρόπο που ε, ε, αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό και όχι από αυτούς που θα καταψηφίσουν. Γιατί στην ουσία υπονομεύεται τα θεσμικά μας όργανα και η νομοθεσία που εμείς πολύ πρόσφατα εγκρίναμε σε, συνδυασμό, σε συνεργασία με άλλους. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο λόγος είναι σε άλλα μέλη. Πρώτα η κυρία Γιούσου. Eh, Πρώτα κυρία Γιούζο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω με όσα είπε ο κύριος Φιέλνερ και θα προσθέσω και κάτι άλλο. Συζητούμε κατά πόσο είναι επιζήμιες για την υγεία ε, ε οι ποικιλίε αυτές και όχι το τι σχέση έχουν με τα φυτοφάρμακα. Το ερώτημα είναι αν είναι ασφαλή για την υγεία και είναι. Αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν θέλω λοιπόν να στηρίξω αυτή την αντίρρηση. Ευχαριστούμε κυρία Κάντεμπαχ. I couldn't disagree more. Εγώ διαφωνώ απολύτως. Διαφωνώ απολύτως. Κοιτάξτε τώρα. Και πολύ σύντομα για, τις, για τους δυο αυτούς, για τα δυο αυτά είδη καλαμποκιού γενετικά τροποποιημένων που είναι ανθεκτικά κατά γλυφοσάτης και γλυφοσινάτης. Και με την έγκριση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος μπορέσαμε να φτιάξουμε την Εξεταστική Επιτροπή για τα ζυζανιοκτώνα, όπου ε, ο στόχος είναι να εξετάσουμε τα επιστημονικά δεδομένα τα οποία συνηγορούν υποτίθεται υπέρ της παράτασης χρήσης της γλυφοσάτης. Και να δούμε από πού βρέθηκαν τα στοιχεία αυτά. Διότι υπάρχει σημαντικό αριθμός ευρωβουλευτών που θεωρούν σημαντικο αριθμό ευρωβουλευτων που θεωρουν οτι η έγκριση χρήσης, η αδειοδότηση δηλαδή της έρχεται σε αντίθεση με την ορθή εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης και ότι εδώ υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν ταιριάζουν στον στη συνολικότερη εικόνα. Τώρα, η έγκριση εισαγωγή δύο ειδών καλαμποκιού που είναι ανθεκτικά ακριβώς σε αυτήν την ε, γλυφοσάτη, το νόημα που θα έχει τελικά θα είναι ότι θα αυξηθεί η χρήση γλυφοσάτης. Θα οδηγήσουν δηλαδή οι εισαγωγέ αυτές σε αύξηση των ποσοτήτων χρησιμοποιούμενης γλυφοσάτης. Πρόκειται για είδη αραβοσίτου ή καλαμουγιού, τα οποία επαναλαμβάνω, θα επιτρέψουν ή θα ευνοήσουν περαιτέρω και αυξημένη χρήση γλυφοσάτης. Γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να επιτραπεί η εισαγωγή αυτών και η καλλιέργεια των δυο ειδών καλαμποκιού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω μια ε, υπόσχεση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Γιούνκερ που ήδη το 2014 μιλούσε για τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με τις αδειοδοτήσεις γενετικών τροποποιημένων οργανισμών. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Όμως σύμφωνα με, τη, με, τις, ε, με διαδικαστικούς κανόνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτή η οποία δίνει την αδειοδότηση. Αυτό το θεωρώ απαράδεκτο. Και ούτε νομίζω ότι ο κ. Γιούνκερ θα βρει τη διαδικασία αυτή δημοκρατική. Έκτοτε βέβαια τίποτε δεν έχει γίνει. Τίποτε δεν έχει αλλάξει. Και όταν ρώτησαν ε, τον, ή ε, την αρμόδια επίτροπο στην Ολομέλεια, είπε το πρόσωπο αυτό, ο Κάιτη, ότι Α, αυτό είναι ατυχές, διότι σε άλλες περιπτώσεις, ναι, θα έπρεπε ε, αυτή τη διαδικασία να ακολουθήσουμε θεωρώ και πάλι ότι ορθώς ο κ. Γιούνκερ θεωρεί μη δημοκρατικέ διαδικασίε αυτέ. Και εγώ εξακολουθώ να τι βρίσκω μη δημοκρατικέ. Ευχαριστώ. Άλλο κανεί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είστε η κυρία Μπρισίκ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου για τα σχόλια τα οποία παρακολουθήσαμε πολύ προσεκτικά εδώ συζητάμε για δύο εγκρίσεις. Η μία για έναν νέο οργανισμό που είναι συσσόρευση ε, γονιδίων και ο άλλος και η άλλη για έναν μοναδικό. Θεωρούμε ότι ε, σωστά εφαρμόσαμε τις εξουσίες που μας έχει δώσει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και θα σας εξηγήσω γιατί οι έλεγχοι γίνονται, όσον αφορά τον, την αξιολόγηση κινδύνου, γίνονται πολύ προσεκτικά και δεν εντοπίστηκε χάσμα δεδομένων. Και άρα υπήρξε συμπέρασμα με βάση την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων και το περιβάλλον. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό, επειδή παρακολούθησα προσεκτικά τα σχόλια, κάποια, κάποιοι, ε, κάποια κράτη σχολίασαν τις αιτήσεις αυτές και η ΕΦΣΑ απάντησε. Το ίδιο ισχύει για τα σχόλια που έγιναν από το, ε, από το κοινό όχι για τον ενιαίο οργανισμό, αλλά για την συσσόρευση των γονιδίων και δεν προσφέρθηκαν νέες πληροφορίες που να ακυρώνει τη θετική άποψη για τον Αραβόστο. Υπό το φως αυτών των πληροφοριών προτείνουμε στα κράτη-μέλη να υπερψηφίσουν και εδώ, κάποια μέλη εδώ είπαν ότι δεν υπάρχει γνωμοδότηση της μόνιμης επιτροπής στις 16 Ιανουαρίου και ως εκ τούτου πρέπει να πάει στην Επιτροπή Θέσεων. Πράγμα που θα συμβεί την ερχόμενη εβδομάδα, 26 Φεβρουαρίου άκουσα πολύ προσεκτικά τις ανησυχίες που αφορούν τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, δηλαδή το γλυφοζάτ και το γλυφοσυνικό αμμόνιο. Έχετε δίκιο, ε, οι, ε, αραβόστοι αυτοί έχουν αντοχή. Οποιοδήποτε, ε, οποιοδήποτε φυτό καλλιεργείται εκτός Ευρώπης, των οποίων το προϊόντα εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να ε, συμμορφώνονται με τα μέγιστα επίπεδα υπολοιμάτων για τα οποία αποφασίζουμε εμείς στην Ευρώπη. Και τα μέγιστα αυτά επίπεδα υπολοιμάτων είτε αφορούν το γλυφοσάτ, το γλυφοσυνικό ή άλλα, τίθενται από εμά και ε, ε, ισχύουν για όλα τα εισαγόμενα προϊόντα περιλαμβανομένων και των τροφών και τροφίμων από γενετικά ε, τροποποιημένους οργανισμούς, και αυτών που συζητώνται σήμερα. Δεν είναι αυτά λοιπόν τα φυτά που θα έρθουν και θα βλάψουν το περιβάλλον ή την ανθρώπινη και υγεία και την υγεία των ζώων. Όλα αυτά τα έχουμε, για όλα αυτά έχουμε νομοθετήσει εμείς. Τώρα όσον αφορά ένα άλλο σκέλος που άκουσα να αναφέρεται επίσης είναι οι επιπτώσεις των ζυζανοκτώρων που δεν λαμβάνεται υπόψη όντως λαμβάνεται υπόψη γιατί αυτές, οι φυτίες ψεκάζονται από το ζυζανιοκτόνο εκτός Ευρώπης και αυτό οδηγεί σε πιθανές αλλαγές στη σύνθεση την φαινοτυπική και ε, τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά και τα αγρονομικά τους χαρακτηριστικά, τα γεωπονικά τους χαρακτηριστικά. Υπάρχει ένα άλλο στοιχείο επί του οποίου σχολιάσατε είναι οι επιπτώσει στη βιοπικιλότητα. Μην, ε, μην ξεχνάμε, μην υποτιμάμε ότι οι χώρες που, που καλλιεργούν αυτούς τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς είναι ε, χώρες ε, ε ανεξάρτητες, και δεν μπορούμε να τους επιβάλλουμε τη μη καλλιέργεια. Ε, εμείς δεν μπορούμε να τους πούμε ε, να μην καλλιεργούν επειδή αυτό είναι δικαίωμά τους. Τέλος, όσον αφορά την ε, αξιολόγηση του συνδυασμού, ε, άκουσα ότι δεν ελέγχεται σωστά. Η ΕΦΣΑ ελέγχει τη συσσόρευση των στοιχείων και και είναι πάρα πολύ δύσκολο να υποστηρίξει κανείς ότι η άποψη του ΕΦΣΑ είναι ανεπαρκής. Είναι πάρα πολύ δύσκολο τουλάχιστον για την Κομισιόν να έχει τα στοιχεία και να πει ότι η, η γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ δεν συνάδει με την νομοθεσία και τις κατευθυντήριες γραμμές. Άκουσα επίσης την έκκληση για περισσότερη δημοκρατία. Έχουμε φυσικά ως Επιτροπή υποβάλει μια πρόταση προς το Συμβούλιο και στο ε, Κοινοβούλιο που, προτείνεται ότι οι, τα κράτη-μέλη να περιορίσουν τις εισαγωγές ε, τροποποιημένων γενετικά τροφών και ε, ζωοτροφών γιατί αυτά τα οποία συζητάμε εισάγονται σήμερα. Έχουμε στείλει μια πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να περιορίσουν τις εισαγωγές τους η οποία απορρίφθηκε ήδη από το Κοινοβούλιο. Τώρα το θέμα της επιτροπολογίας Τουρκίας προτείνατε ότι θα πρέπει να απορριφθούν όλες οι προτάσεις επί, το οποίο, επί των οποίων δεν υπάρχει γνωμοδότηση από τη Μόνιμη Επιτροπή. Υπάρχει μια πρόταση της Κομισιόν που εισάγει περισσότερη δημοκρατία και θα θέλουμε να ζητήσουμε από εσά και συνολικά από το Κοινοβούλιο να ξεκινήσετε μια συζήτηση και να τροφοδοτήσετε θετικές συζητήσεις και να εμπλέξετε και το Συμβούλιο ώστε να υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσμα της επιδίωξης για περισσότερες δημοκρατίες. Εν κατακλείδη μπορώ να πω ότι η Κομισιόν δεν έχει λόγο λόγο να αποσύρει αυτές τις γνωμοδοτήσεις, τις αποφάσεις. Καταρχήν τα θέματα του, επί των οποίων ρωτά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν σχέση με αυτά, αλλά και στο παρελθόν και σήμερα είμαστε διαθέσιμοι να απαντήσουμε σε όλα σας τα ερωτήματα και ελπίζουμε ότι τουλάχιστον έχουμε ε, απαντήσει σε κάποιες από τις ανησυχίες σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η συζήτηση για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Ε, η ψηφοφορία θα γίνει του ε, αύριο. Αυτά για σήμερα. Υπάρχει μερίσια διάταξη για αύριο. Έχει εγκριθεί. Θα, θα τα πούμε αύριο. 9 η ώρα είναι συνεδρία των συντονιστών και 10 και 4 για τα μέλη της Επιτροπής. Καλό σας βράδυ.